Mesdames et messieurs, je vous invite à prendre... Με μεγάλη χαρά θα καλωσορίσω τη Βαρόνια Άστον. Κυρία Κάθρι Άστον είναι ύπατη εκπρόσωπος Ευρωπαϊκής Ένωσης για Εξωτερικές Υποθέσεις και Θέματα Ασφαλείας και Αντιπρόεδρος τη Ευρωπαϊκής Επιτροπής σύμφωνα με τη δέσμευση που είχε αναλάβει να έρχεται μια φορά το χρόνο στην Επιτροπή μας. Είναι η δεύτερη φορά που μας επισκέπτεται για μια ανταλλαγή απόψεων. Εν τω μεταξύ έγιναν πολλά πράγματα από την τελευταία συνάντηση. Η θέση σε λειτουργία της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης, η υπηρεσία της οποίας οι μέθοδοι εργασίας ενεκρίθησαν και από τη Γενική Διεύθυνση ΔΕΦΚΟ της Επιτροπής. Πρόσφατα το Κοινοβούλιο δέχτηκε νέες προτάσεις για νέες μεθόδους χρηματοδότησης στα πλαίσια του προγραμματισμού των νέων μέσων για την χρηματοδότηση της συνεργασίας για την ανάπτυξη, η νομοθετική πρόταση περιλαμβάνει πολλές τροποποιήσεις, οι οποίες δεν είναι διόλου ανώδυνες, όπως η μείωση της συνεργασίας για την ανάπτυξη με τις αναδυόμενες χώρες ή η δυνατοτητα από κοινού προγραμματισμού με τα κράτη-μέλη. Η κυρία Αστόν είναι μαζί μας λοιπόν, την ευχαριστώ για μια ακόμη φορά και θα μας δώσει τη δική της αντίληψη για τον τρόπο με τον οποίο θα προχωρήσουμε στην ενσωμάτωση της πολιτικής της αυτής της γενικότερες πολιτικές της Ένωσης. Χωρίς άλλη καθυστέρηση θα δώσω το λόγο στη Λεδιάστον. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Έχουμε καιρό να τα πούμε, λέει η Βαρόνη. Και ένα από τα πράγματα τα οποία ελπίζω να μπορέσουμε να συζητήσουμε κατά τη διάρκεια της συνάντησης αυτής είναι να μπορέσετε να συνεισφέρετε πολιτικά. Είναι σημαντική η άποψή σας και περιμένω τις απόψεις σας για τον τρόπο με τον οποίο θα εφαρμόσουμε τις πολιτικές μας. Είμαι σε συζήτηση με την Προεδρία της Δανίας και την Προεδρία της Κύπρου για να δούμε τι άλλο μπορούμε να κάνουμε έτσι ώστε η Επιτροπή μας να μπορέσει να συνεισφέρει και αυτή όσο μπορεί. Εν πάση περιπτώσει με μεγάλη χαρά παίρνω το λόγο. Η χρονιά την οποία περάσαμε ήταν προκλητική. Η Αραβική Άνοιξη, Πράγματι κυριάρχησε της πολιτικής μας στη γειτονία και η ευρωπαϊκή οικονομική κρίση και αυτή ήταν, ήταν κάτι το οποίο εν πολλής έδωσε μια νέα εικόνα για την κατάσταση. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι κάτω από αυτές τις δύσκολες οικονομικά συνθήκες και στα πλαίσια των αλλαγών που διαπιστώνουμε στον κόσμο, η εκρίζωση της ένδυας και η αηφορία στην ανάπτυξη είναι πολιτικές οι οποίες παραμένουν σημαντικές και θα γίνουν σημαντικότερες. Οι πολιτικές αυτές ε, πρέπει να παραμείνουν, θα έλεγα, στο κέντρο της ανησυχίας της Ένωσης. Έχει υπάρξει σίγουρα μια κάποια πρόοδος στον τομέα της ε, εκπαίδευσης. 9 εκατομμύρια παιδιά εντάχθηκαν σε συστήματα παιδείας, 5 εκατομμύρια παιδιά εμβολιάστηκαν για μαγουλάδες σαν παράδειγμα, ε, και επίσης χιλιάδες κόσμος έτυχε θεραπείας ε, με φροντίδα της Ένωσης ε, για το AIDS. Συνολικά επηρεάσαμε σχεδόν 50 εκατομμύρια κόσμο θετικά και υπάρχουν πολλοί τρόποι επιρροής, ιδιαίτερα στην κοινωνία των πολιτών. Από την αρχή της Αραβικής Άνοιξης βλέπουμε ότι υπάρχουν χώρες οι οποίες έχουν φτάσει σε ένα αποφασιστικό σημείο της μεταβατικής διαδικασίας Στόχος μας είναι όσο προχωρούν η δημιουργία των θεσμών, η δημιουργία του τρόπου με τον οποίο θα στηρίξουν τους πληθυσμούς τους οι χώρες αυτές, τα πολιτικά προγράμματα τα οποία θα πρέπει να διασφαλίσουν η δημοκρατία, η ελευθερία, τα ανθρώπινα δικαιώματα, η ισότητα, η έννοια του να κερδίσει κανείς από μια διαδικασία η οποία πρέπει να είναι παραγωγική. Αυτό συνδεδεμένο με την οικονομική ανάπτυξη και με την αηφόρο ανάπτυξη είναι κάτι το οποίο είναι απαραίτητο έτσι ώστε κάθε κοινωνία να μπορέσει να ωφεληθεί. Πολιτικές στον τομέα της παιδείας, πολιτικές κοινωνικές στον τομέα της καταπολέμησης της φτώχειας, όλα αυτά θα πρέπει να υποστηριχθούν με συγκεκριμένο τρόπο. Η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη, προκλητικά δύσκολη και όχι μόνο στις χώρες της γειτονίας αλλά και πέραν αυτών. Όταν βλέπει κανείς τον τρόπο με τον οποίο αλλάζουν τα πράγματα στην υποσαχαρική Αφρική σαν παράδειγμα και όταν βλέπει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν χώρες ε, πέραν ε, της Ευρώπης, ε, δηλαδή στην Καραϊβική, στον Ειρηνικό κτλ. Πρέπει να υπάρξει νέα πολιτική δυναμική έτσι ώστε οι επιπτώσεις θα έλεγα της Αραβικής Άνοιξης να είναι θετικές. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε να προλάβουμε δυσάρεστες καταστάσεις και θα πρέπει να μην χρησιμοποιηθούν οι αλλαγές αυτές για πιο κατασταλτικές πολιτικές. Υπάρχουν προβλήματα και στα πλαίσια της αηφόρου αναπτύξεως λόγω των κλιματολογικών αλλαγών. Πρέπει οι στόχοι για την εκρίζωση της φτώχειας να συνεχίσουν να είναι μπροστά μας και να στηρίζουμε τις χώρες που πολεμούν να τους πετύχουν με συγκεκριμένο τρόπο. Τον 21ο αιώνα δεν πρέπει να μιλάμε για λοιμούς στον κόσμο μια από τις πραγματικές τραγωδίες που αντιμετωπίζουμε. Δυστυχώς το 2012 έχουμε τέτοια προβλήματα, πρέπει να βρούμε στρατηγικές για να αντιμετωπίσουμε τους λοιμούς, πρέπει να βρούμε βραχυπρόθεσμα μέσα αντιμετώπισης τους και όχι μακροπρόθεσμα, δυστυχώς. Αυτό που μπορώ να πω λοιπόν είναι ότι αν δει τα πράγματα καλά τη στρατηγική μας μετά τη Λισαβόνα, μετά τη συνθήκη τη νέα, βλέπουμε ότι και πά και η αναπτυξιακή πολιτική θα πρέπει να συνδεθούν με ένα σωστό τρόπο. Η ασφάλεια για τους πολίτες δεν είναι μόνο κάποια κρίσιμα θέματα που αφορούν την αποτροπή του πολέμου και των ένοπλων συγκρούσεων, αλλά είναι η ασφάλεια στην προμήθεια τροφίμων, είναι η αντιμετώπιση των κλιματολογικών αλλαγών, είναι η ζωή σε μια κοινωνία που παρέχει ένα δίκτυο ασφαλείας και κυβερνήσεις που μπορούν να βοηθήσουν τους πληθυσμούς τους. Γι' αυτό και αναπτύσσουμε τις στρατηγικές αυτές και στην περιοχή του Σαχέλ. Προσπαθήσαμε να έρθουμε σε επαφή με τους υπουργούς εξωτερικών όλων αυτών των χωρών. Προσπαθήσαμε να συνεργαστούμε μαζί τους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Συνεργαζόμαστε και με την κοινωνία των πολιτών στις περιοχές αυτές έτσι ώστε να καταλήξουμε σε στρατηγικές οι οποίες συνολικά θα μας επιτρέψουν τη διασφάλιση της ασφάλειας σε όλους τους τομείς που είπα. Μακράν των λιμών λοιπόν, μακράν αυτών οι οποίοι θέλουν να στρατολογήσουν νέα παιδιά και να τα κάνουν τρομοκράτες, υποστήριξη των μικρών κοινοτήτων και των χωριών που πιστεύουν ότι υπάρχει δυνατότητα να αποδείξουν οι κυβερνήσεις τους ότι θα τους βοηθήσουν. Σαν παράδειγμα μικρές κλινικές στον τομέα της υγείας, κάτι το οποίο θα βοηθήσει και τις αδυνάμεις ασφαλείας να λειτουργήσουν σωστά, να μπορέσουν να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας, να μπορέσουν να στηρίξουν την οικονομική ανάπτυξη και να στηρίξουν και την κοινωνία των πολιτών την ίδια έτσι ώστε αυτή με τη σειρά της να λειτουργήσει υποστηρικτικά στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να συγκεντρώσουν την προσοχή τους στο είδος της διακυβέρνησης η οποία είναι κατάλληλη για την χώρα και την περιοχή. Ε, με τους συναδέλφους μου συνεργάζομαι πολύ καλά, όπως με τον άντρο Σπίτβαλτς, αλλά και με άλλους επιτρόπους όπου καλύπτουμε περιοχές του κόσμου οι οποίες αντιμετωπίζονται από έκτακτες κρίσεις, Πακιστάν, η Ιαπωνία με το τσουνάμι και χώρες οι οποίες αντιμετωπίζουν τρομερές ε, ανατάραχες όπως η Εμένη που προσπαθήσαμε να διασφαλίσουμε την παρουσία των τροφίμων στην περιοχή και προσπαθήσαμε και μακροπρόθεσμα και βραχυπρόθεσμα να λειτουργήσουμε θετικά. Υπάρχουν χώρες τις οποίες πρέπει να εμπλακούμε όπως το Νότιο Σουδάν γιατί υπάρχουν πάρα πολλές δυσκολίες, τις οποίες ίσως θα αναφερθούμε αργότερα. Πρέπει να αναπτύξουμε ένα πνεύμα συνεργασίας ανάμεσα στα όργανα της Ένωσης. Είναι κάτι το οποίο επιθυμούμε όλοι και έχουμε όλοι επενδύσει σε αυτό. Δεν υποκρίνομαι ότι δεν υπάρχουν δρόμοι που δεν έχουμε δοκιμάσει. Παρ' αυτά έχουμε μια νέα υπηρεσία στη διάθεσή μας και έτσι μπορεί ίσως να βρεθούν και νέοι τρόποι συνεργασίας. Νέοι τρόποι οι οποίοι θα μας εξασφαλίζουν ότι θα λειτουργούμε συνεκτικά και συνολικά. Θα πρέπει εδώ να τιμήσω και να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους και στην ΤΕΦΚΟ και στην Γενική Διεύθυνση Εμπορίου και στη Γενική Διεύθυνση ε, διαχείρισης κρίσεων και στη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος και στη δική μου υπηρεσία για τον τρόπο με τον οποίο συνεργάζονται. Ο στόχος μας είναι να υπογραμμίσουμε σωστά τους στόχους της ε, τήρησης της τάξης, των οικονομικών προοπτικών και τη συνεργασία σε εταιρική βάση. Είπα ότι οι προκλήσεις είναι τεράστιες. Γνωρίζετε όμως ήδη ότι προσπαθούμε να δημιουργήσουμε τις συνθήκες έτσι ώστε αυτά τα οποία να κάνουμε να προλαμβάνουν κοινωνικές αναταράξεις οι οποίες θα δημιουργήσουν με τη σειρά του σοβαρά προβλήματα στον κόσμο. Αυτοί οι οποίοι βρίσκονται πολλές φορές σε περιοχές ε, ε, με συγκρούσεις οδηγούν στα παιδιά να εγκαταλείπουν φυσικά την εκπαίδευση, ε, σε αδυναμία ανάπτυξης της οικονομίας, και φυσικά η βία καταστρέφει τους ανθρώπινους ε, ιστούς, τους κοινωνικούς ιστούς, τους οποίους τόσο έχουν ανάγκη οι άνθρωποι. Απαιτείται να υπάρξει σε αυτές τις περιοχές αναπτυξιακή βοήθεια, αλλά και βοήθεια στον τομέα της στήρησης της ηρεμίας και της ειρήνης. Ένα παράδειγμα που δείχνει πόσο έχουμε προχωρήσει τα τελευταία χρόνια είναι στο κέρας της Αφρικής έχουμε μία στάση εκεί η οποία καλύπτει πολλούς τομείς ταυτόχρονα. Έχουμε σαν παράδειγμα ε, τρόπους αντιμετώπισης του φαινομένου της πειρατείας. Προσπαθούμε να ελαφρύνουμε τους φόβους αυτών οι οποίοι εμπορεύονται στην περιοχή. Υπάρχουν πάρα πολλές χώρες του κόσμου που πηγαίνουν εκεί για εμπορικούς λόγους αλλά φοβούνται ότι θα υποστούν επιθέσεις, πειρατεία από πολλούς οι οποίοι ε, εμπλέκονται σε παράνομες δραστηριότητες. Προσπαθούμε να δούμε ε, τις συνέπειες που έχει στην οικονομία της περιοχής αυτής τέτοιες δραστηριότητες, εμποδίζουν την ανάπτυξη την οικονομική, εμποδίζουν τον τουρισμό και ταυτόχρονα θα πρέπει το Παγκόσμιο Πρόγραμμα Τροφίμων να διασφαλίσει την παροχή τροφίμων στις πιο φτωχές περιοχές του κόσμου. Έχουμε αυτή τη στιγμή πέντε στρατιωτικά σκάφη ανοιχτά των ακτών του κέρατος της Αφρικής και πολύ συχνά έχουμε και άνω των 10 για να διασφαλίσουν την ασφάλεια και την ανάπτυξη της περιοχής. Όταν επισκέπτεται Κανείς βέβαια τους, ε, ε, τους υπεύθυνους των στρατιωτικών αυτών σκαφών ε, σου λένε ότι το πρόβλημα πρέπει να αντιμετωπιστεί στη ρίζα του, πρέπει να αντιμετωπιστεί δηλαδή στην ενδοχώρα. Γιατί εκεί πολύ συχνά νέοι άνθρωποι, πολλοί, πολλά, πολλοί νέοι άνθρωποι, παιδιά σχεδόν, δελεάζονται με χιλιάδες δολάρια για να εμπλακούν σε εγκληματικές δραστηριότητες. Πρέπει λοιπόν η πολιτική μας και η στρατηγική μας να είναι συντονισμένη και αυτό θα πρέπει να γίνεται με τη στήριξη των ηγετικών κατηγοριών της περιοχής στο Σόμαλιλάν, στο Πούντλαντ, τους λαούς της περιοχής, Τανζανία, Κένια, Σεϊχέλες, Μαυρίκιος, όλες αυτές οι χώρες πρέπει να συνεργαστούν έτσι ώστε να υπάρξει μια λύση και μπορούμε να συνεργαστούμε μαζί τους. Μια πολιτική λύση μια ανάπτυξη των ανθρωπιστικών προγραμμάτων και μια προσπάθεια έτσι ώστε να αποτρέψουμε την πειρατεία εις βάρος των εμπορικών πλοίων και να διασφαλίσουμε την, την αυθονία τροφίμων για τους πληθυσμούς της περιοχής. Όταν μιλάει κανείς για την ευημερία των κατοίκων των περιοχών πρέπει να δούμε τι ρόλο μπορούμε να παίξουμε στα πλαίσια και των χωρών ΑΚΕ και μαζί με τις χώρες ΑΚΕ. Ξέρω και ξέρετε κι εσείς τον τρόπο με τον οποίο συνεργαζόμαστε με τις χώρες ΑΚΕ. Αφρική, Καραϊβική, Ειρηνικός. Πρέπει λοιπόν να εντατικοποιήσουμε τις σχέσεις μας. Ξέρετε ότι η υπηρεσία μου έχει προχωρήσει σε, προγραμματικά, ε, σε προγραμματικές περιόδους ήδη από το 2011 συνεργασίας με τις χώρες ΣΑΚΕ. Εδώ και η δική σας συνεισφορά από πλευράς του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ήταν θετική. Και η αντιπρόεδρος της ε, ε, Μικτής Κοινοβουλευτικής, ε, ΕΟΚΑΚΕ, Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΚΕ, είναι σημαντική. Η εμπειρογνωμοσύνη την οποία έχετε είναι για μας καθοριστική, έτσι ώστε να ορίσουμε σωστά τις ανάγκες των προγραμμάτων και έτσι ώστε να μπορέσουμε να τηρήσουμε μία στάση θα έλεγα απέναντι στα προβλήματα η οποία να είναι κυρίαρχα αναπτυξιακή, ε, να στηρίξουμε την αηφορία, να στηρίξουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία. Όταν βλέπουμε τις αλλαγές οι οποίες θα πρέπει να γίνουν, και ξέρω ότι τα έχετε συζητήσει αυτά και με τον Άντερ Σπίμπαλς, ο οποίος είναι πρωτοπόρος θα έλεγα, στον τρόπο με τον οποίο χορηγείται η βοήθεια, έτσι ώστε η βοήθεια αυτή να φτάνει στους δικαιούχους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και προσπαθούμε η βοήθειά μας να είναι όσο περισσότερο γίνεται αποτελεσματική, αναγνωρίζοντας ότι οι φτωχότεροι πολλές φορές δεν είναι στις φτωχότερες χώρες οι φτωχότεροι μπορεί να ζουν σε χώρες τις οποίες θα μπορούσαμε να περιγράψουμε χώρες μεσαίου εισοδήματος. Έτσι όπως προχωρούμε και αναπτύσσουμε τις σχέσεις μας με τις χώρες αυτές, πρέπει να τις καταστήσουμε ικανές να έχουν στη διάθεσή τους τα κατάλληλα προγράμματα που θα φροντίσουν τους φτωχότερους των κοινωνιών τους. Αυτό είναι ιδιαίτερα κρίσιμο για τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε εμείς τη δουλειά μας. Αυτό είναι ένα κομβικό κομμάτι της εταιρική σχέσης που έχουμε μαζί τους. Αυτό δεν συμβαίνει πάντα. Πάρα πολλές φορές υπάρχουν πολιτικοί λόγοι για τους οποίους αυτοί που έχουν χρήματα θέλουν να τα κρατήσουν και δεν θέλουν να επηρεάσουν θετικά. Πάρα πολύ συχνά έχει άμεση σχέση η υπόθεση αυτή με την ανικανότητα των κρατικών θεσμών να μπορέσουν να είναι αποτελεσματικοί επιτόπου. Πρέπει λοιπόν όλα αυτά συνολικά να τα δούμε έτσι ώστε να βοηθήσουμε κάποιες κοινότητες οι οποίες είναι ίσως πτωχές και αγροτικές καθαρά να αναπτυχθούν, να βελτιώσουμε τις διαδικασίες δημιουργίας υποδομών, να στηρίξουμε την τοπική οικονομία, να στηρίξουμε τα τοπικά συστήματα εκπαίδευσης για τους νέους φυσικά, να μπορέσουμε να τους βοηθήσουμε έτσι ώστε να διαθέσουν τα προϊόντα τους στις αγορές με αποτελεσματικό τρόπο. Τα είδα όλα αυτά πολύ αποτελεσματικά στην IT. Εκεί βλέπει κανείς το, τι χρειάζεται να γίνει στα διαφορετικά σημεία της νήσου αυτής έτσι ώστε να στηρίξουμε τους κατοίκους της να τους καταστήσουμε ικανούς σε επίπεδο γεωργικό, να αναπτυχθούν πέραν του απλά να παράγουν για εξαγωγή, να τους βοηθήσουμε να επεξεργάζονται τα προϊόντα τους, να τους βοηθήσουμε να δώσουν εκπαιδευτικές δυνατότητες στους νέους τους και να μπορέσουν να δημιουργήσουν προϊόντα, νέα προϊόντα και να μπορέσουν να διαχειριστούν την παραγωγή τους και να ενταχθούν στην συνολική διαδικασία επεξεργασίας και εμπορίας των προϊόντων τους. Λοιπόν, υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα δεν θα καθυστερήσω πολύ γιατί θέλω να περάσω στο πιο σημαντικό κομμάτι της συνάντησής μας που είναι οι ερωταπαντήσεις. Αλλά πολλές φορές κάποιες από αυτές τις χώρες προσπαθούν, κάνουν καλά πράγματα αλλά δεν βοηθούνται οι κοινωνίες τους να αναπτυχθούν σωστά. Το θέμα δεν είναι να τους δίνουμε βοήθεια. Είναι μια φιλοσοφική στάση αυτή, η οποία από πάνω προς τα κάτω δεν βοηθάει. Το θέμα είναι από κάτω να βοηθήσουμε. Να πρέπει να τα προγράμματα τα οποία προχωράμε και εφαρμόζουμε να δώσουν τις δυνατότητες στους πολίτες τους ίδιους να αναπτύξουν τα προγράμματά τους και να αναπτυχθούν με τη σειρά τους. Κάποιες από τις χώρες με τις οποίες συνεργαζόμαστε είναι στρατη, στρατηγικοί εταίροι είναι χώρες άλλες με τις οποίες τώρα ξεκινούμε να συνεργαζόμεθα. Είναι χώρες οι οποίες τώρα έχουν αρχίσει να βελτιώνουν τις συνθήκες για τους πληθυσμούς τους, έτσι ώστε οι πληθυσμοί τους να αποφασίζουν για το μέλλον τους. Τώρα, λίγα πράγματα για τις κλιματολογικές αλλαγές. Αυτό είναι ένα συγκεκριμένο θέμα, το οποίο πρέπει να μας απασχολήσει στον τομέα της αηφορίας της ανάπτυξης είναι αλήθεια και πρόβλημα για μικρές χώρες, ιδιαίτερα για μικρές νησιωτικές χώρες, χώρες νήσου στην Καραϊβική και στον Ειρηνικό. Μέλη της Επιτροπής σας είδαν τις επιπτώσεις της κατάστασης σε κάποιες τέτοιες χώρες περιοχές. Πρέπει λοιπόν να το αντιμετωπίσουμε συνολικά το θέμα. Πρέπει να συνεργαστούμε με τους επιτρόπους οι οποίοι ασχολούνται ειδικά με τα θέματα. Πρώτον, μετριάζοντας τις συνέπειες της αρνητικές των κλιματολογικών αλλαγών σήμερα και στο μέλλον, Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί για τον τρόπο με τον οποίο θα υποστηρίξουμε τις χώρες οι οποίες λόγω των κλιματολογικών αλλαγών πρέπει να κάνουν ορισμένα πράγματα με διαφορετικό τρόπο. Βλέπουμε ότι υπάρχουν χωριά που καταστρέφονται σχεδόν κάθε χρόνο από τις πλημμύρες. Πώς θα στηρίξουμε τις περιοχές αυτές για να μην καταστρέφονται πλέον και πώς θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε τις κοινότητες αυτές να κρατήσουν αυτά τα οποία για αυτούς είναι σημαντικά. Πρέπει λοιπόν να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τις κοινότητες να χρησιμοποιήσουν τις νέες συνθήκες που δημιουργούνται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Πρέπει να συνδέσουμε τις στρατηγικές μας παρεμβάσεις, οι οποίες είναι μεγάλες αξίες θα έλεγα και στόχοι, σε σχέση με τις κλιματολογικές αλλαγές, αλλά να πάρουμε και μέρος μακροπρόθεσμα σαν πρωταγωνιστές στην αντιμετώπιση των προβλημάτων και την έβρεση των λύσεων σε όλο τον κόσμο. Εδώ η ανάπτυξη είναι απαραίτητη. Λίγα λόγια τώρα για το Σουδάν, το νότιο Σουδάν. Εγώ είμαι σε επαφή και την ηγεσία και των δύο χωρών. Είπα στον πρόεδρο του Νοτιού Σουδάν όταν συναντήθηκα μαζί του ότι ήμουν πολύ περήφανη που ήμουν μια πάρα πολύ ζεστή μέρα να σηκώνεται για πρώτη φορά η σημαία αυτής της χώρας. Μια χώρα όμως πάρα πολύ εύθραστη. Μια νέα χώρα η οποία πρέπει να υποστηριχθεί όσο γίνεται καλύτερα και σε επίπεδο αναπτυξιακών δυνατοτήτων και σε επίπεδο δημιουργίας και κατασκευής υποδομών που είναι πάρα πολύ ισχνές, αλλά και σε επίπεδο συνεργασίας με τα κράτη-μέλη. Στην Τζούμπα, στην ουσία, ε, όλες οι οργανώσεις, ε, θα έλεγα, βοήθεια, συνεργασίας κτλ και οι διπλωματικοί εκπρόσωποι είναι στην ίδια περιοχή, στον ίδιο χώρο. Πρέπει λοιπόν να συνεργαστούμε στενά για να βοηθήσουμε τη χώρα αυτή. Σαν παράδειγμα το νέο αεροδρόμιο. Ε, πρέπει να μπορέσουν να προχωρήσουν, πρέπει να μπορέσουν να λύσουν τα προβλήματα που έχουν με το Βόρειο Σουδάν. Πρέπει να στηρίξουμε αυτά τα οποία κάνει ο πρόεδρος Σουμπέκη. Ε, πρέπει να τους βοηθήσουμε να βρουν μια λύση για τον αγωγό γιατί είναι πολύ σημαντικός για την οικονομία τους. Πρέπει να βρουν τρόπους να βρουν ποικίλε μορφές προσόδου για την οικονομία τους, έτσι ώστε να εκμεταλλευτούν όλες τις δυνατότητες της χώρας τους. Λοιπόν, ξέρετε ότι τον Απρίλιο έχει συμφωνηθεί με τη Σαν Γιουκή να πάω στη Βυρμανία και ο Άντερς Πιμπάλς την έχει ήδη συναντήσει και προσπαθούμε να δημιουργήσουμε επαφές όπου αυτές είναι απαραίτητες. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι έχουμε σαφέστατες προσδοκίες για την Βυρμανία. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι οι εκλογές θα πάνε καλά, ότι οι υπόλοιποι πολιτικοί κρατούμενοι θα απελευθερωθούν, ότι πρέπει να υπάρχει πλήρης ανθρωπιστική πρόσβαση στην περιοχή και ότι πρέπει παράλληλα να τελειώσουν οι σειράξεις οι περιφερειακές. Εύχομαι ότι πρέπει να στηριχθούν όλοι αυτοί οι οποίοι εργάζονται για την αλλαγή της πολιτικής κατάστασης και της δημοκρατίας στην βιρμανια Μιανμάρ και ελπίζω ότι όταν πάμε εκεί θα έχουμε μια ξεκάθαρη ευρωπαϊκή πολιτική και συνεκτική ευρωπαϊκή πολιτική. Θα μπορούσα να μιλήσω για πάρα πολλά μέρη του κόσμου, για το Αφγανιστάν με πολλές λεπτομέρειες να αναφερθώ στην εξαιρετική δουλειά η οποία γίνεται στο σύνολο της Αφρικής από τις αντιπροσωπείες μας, οι οποίες συνεργάζονται ε, με τις διευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και με τις πρεσβείες των κρατών μελών. Δύο πράγματα θέλω να πετύχω. Καταρχάς, μια μεγαλύτερη συνεκτικότητα ανάμεσα στα όργανα, τα θεσμικά και τα κράτη-μέλη από την άλλη, έτσι ώστε τα χρήματά μας για την ανάπτυξη να αποδίδουν περισσότερο από όσο σήμερα. Να κάνουμε τις οικονομίες κλίμακας εκεί που χρειάζεται και να προσπαθήσουμε με αυτόν τον τρόπο να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα με ενιαίο τρόπο, με συντονισμένο τρόπο. Θα πρέπει επίσης να προσπαθήσουμε να το πετύχουμε αυτό σε εταιρική σχέση με όλες τις χώρες οι οποίες, ε, στις οποίες εμπλεκόμεθα, σε συνεργασία με τις διεθνείς οργανώσεις όπως τα Ηνωμένα Έθνη και σε συνεργασία φυσικά και με σας. Αυτό έχει σημασία και για το Ευρώπη 2020 και για τους γενικότερους πολιτικούς μας στόχους. Ένα παράδειγμα εδώ για να καταλάβετε πόσο σημαντικό είναι αυτό που κάνουμε. Προσπαθούμε την δουλειά την οποία κάνουμε να τη συνδέσουμε με την προσπάθεια θα έλεγα να υπάρξουν επενδύσεις από τον ιδιωτικό τομέα στις χώρες αυτές. Να πείσουμε και τις διεθνείς επενδυτικές δομές όπως η Παγκόσμια Τράπεζα, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, η Ευρωπαϊκή Επενδυτική Τράπεζα να βοηθήσουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε χώρες μετάβασης όπως λέμε. Σε χώρες οι οποίες ε, μπορεί να φτάσουν να αντιπροσωπεύουν αυτό που εμείς αντιπροσωπεύουμε σήμερα σε οικονομικό επίπεδο στη διεθνή σκηνή. Κάποιες από τις χώρες αυτές τώρα ξεκινούν τις διαδικασίες. Τώρα εδώ βρίσκομαι ανάμεσα σε κοινοβουλευτικού εκπροσώπους και θέλω να τους ευχαριστήσω για τη συνεισφορά τους όταν συνεργάζομαι μαζί τους σε ταξίδια στον κόσμο ε, τους ε, εκτιμούν ιδιαίτερα και γενικά η συμμετοχή σας είναι πολύ σημαντική σε σχέση με την παροχή βοήθειας και σε σχέση με τη σωστή χρήση της βοήθειας. Λοιπόν, θα πρέπει να πείσουμε σε όλες αυτές τις χώρες, όλες αυτές τις χώρες πόσο σημαντική είναι η δημοκρατία, να ικανοποιήσουμε αυτούς οι οποίοι θέλουν να ασχοληθούν με την πολιτική Είχα πάει σε μια συνάντηση 300 γυναικών σαν παράδειγμα στην Λιβύη με φιλόδοξους πολιτικά νέους ανθρώπους στην Τινησία, στην Αίγυπτο, αλλού. Όλες οι χώρες αυτές περνούν μέσα από σημαντικές αλλαγές. Η προσπάθεια που γίνεται από τη μεικτή κοινοβουλευτική και από τις κοινοβουλευτικές σχέσεις μας γενικότερα είναι πολύτιμη δουλειά. Δεν πρέπει να την υποτιμάμε σαν βουλευτές αλλά και γενικότερα και εγώ προσεκτικά θα έλεγα η δουλειά σας ότι όχι μόνο ε, είναι σεβαστή αλλά έχει και αποτελέσματα. Σας ευχαριστώ γι' αυτό. Merci beaucoup, euh, Lady Ashton. Nous allons Ευχαριστώ θερμά, Lady Ashton. Και τώρα το λόγο μπορούν να λάβουν οι συνάδελφοι. Ξέρετε, έχουμε περιορισμού έχουμε και τις ε, ψηφοφορίες άλλωστε μετά. Περιοριζόμαστε λοιπόν στα 2,5 λεπτά ομιλία. Θα ακούσουμε ε, ανά ερωτήσεις, γιατί έχουν υποβληθεί αρκετέ ε, για να έχετε περιθώριο και, και, η Λεδιά να απαντήσει. Ο κύριο Γκάι Μίτσουλ. Πρόεδρε, καλημέρα σας, καλημέρα σας κυρία Άστον και ευχαριστώ ιδιαίτερως για την υποστήριξη που προσφέρει εντυπωσιακή σήμερα η υπηρεσία εξωτερικής δράσης και ελπίζω να συνεχίσει και στο μέλλον. Για, τις, ε, για την ερώτηση μου τώρα. Έχουμε τους στόχους ε, της χιλιετίας. Ερωτώ όμως για την ανάπτυξη συγκεκριμένα πώς μπορείτε να προσμετρήσετε την επίτευξη των στόχων και πόσο συνέπεια ή συνοχή μπορούμε να έχουμε. 30 δισεκατομμύρια για περισσότερη συνοχή θα μπορούσαμε να έχουμε. Μπορείτε να μας σχολιάσετε. Επίσης, στα Φίτζι, στα νησιά Φίτζι, εμείς ως δεύτερος μεγαλύτερος χορηγός, πόσο αντιδρούμε στις εξελίξεις εκεί, Για δε την κατάσταση των μειονοτήτων στη Συρία θα ήθελα να ρωτήσω, γιατί έχουμε ειρηνικές ε, μειονότητες εκεί, ε, ειρηνικές ε, θρησκευτικές μειονότητες που ε, δεν ξέρουμε τι ε, τους επιφυλάσσει η μοίρα. Στην Ιγυρία επίσης οι χριστιανοί έχουν ε, υποστεί επιθέσεις πολύ ενισχυτικές, ιδίως από τα όσα είδαμε και χθες τις ειδήσει. Θα ήθελα λοιπόν να σας παρακαλέσω, μια και δεν θα μπορούσα να συνεχίσω, κάποια σχόλια σε αυτά τα θέματα. Και επίσης, εν παρόδο, και είναι ένα θέμα που με ενδιαφέρει εν γέννη. Ξέρουμε ότι συνήθως ε, σας αποκαλούμε, είπατε εκπρόσωπος ε, και ε, επικεφαλής υπηρεσίας εξωτερικής δράσης Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εγώ νομίζω ότι θα ήταν καλό να σας ονομάσουμε κάτι σαν εκπρόσωπος των εξωτερικών. Ένα τίτλο πιο συγκεκριμένο για να καταλαβαίνει και ο κόσμος τι κάνετε, όχι όλο αυτό το μακρινάρι. Ευχαριστώ κύριε Μίτσελ. Ο κύριος Κόρτης Λάστρα. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Χαίρομαι κυρία Άστον γιατί σας βλέπω εδώ στην Επιτροπή μας. Είναι θα ήταν καλό να είχαμε τέτοιου είδου ανταλλαγή απόψεων περισσότερο συχνά. Αυτό θα εμπλούτιζε τις εργασίες της Επιτροπής μας και θα έδειχνε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει περισσότερη σημασία στα ζητήματα αυτά. Μπορούμε να δουλέψουμε ικανοποιητικά και να καταφέρουμε να εξαλείψουμε τη φτώχεια. Ως προς το DCI, ε, σίγουρα θα έχετε τη στήριξή μας στις διαπραγματεύσεις. Αυτό το πιστεύω. Ωστόσο, θα πρέπει να διατηρηθεί τουλάχιστον το τωρινό επίπεδο χρηματοδότησης. Δεν θα πρέπει η κρίση αυτή ουσιαστικά να μετατραπεί σε δίμιο της ε, ε, πολιτικής, της ευρωπαϊκής πολιτικής στο διεθνές στερέωμα. Η πολιτική μας ομάδα στηρίζει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θέλουμε να έχουμε διαφοροποιημένη βοήθεια και να αφιερώνεται η βοήθεια αυτή σε συγκεκριμένα θέματα, αλλά όχι με οποιοδήποτε τίμημα. Πάντοτε υπό το πρίσμα του στόχου της εξάλληψης της ε, φτώχειας και της θεσμοθέτησης πολιτικών συνεργασίας. Ως πολιτική ομάδα είμαστε ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένοι. Θέλουμε μια αποτελεσματική βοήθεια. Επομένως, η επιδίωξη των στόχων της χιλιετίας είναι βασική σημασίας για την εξάλληψη της φτώχειας. Θέλουμε να δεσμευθείτε ενώπιόν μας ε, ότι θα καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια ε, για την επίτευξη ε, των στόχων της χιλιετίας και να τοποθετηθείτε επί των στόχων μετά το 2015. Στον κόσμο μας σήμερα όλο και περισσότερη φτώχεια επικρατεί, όλο και περισσότερες ανισότητες σημειώνονται, όχι μόνο στην Αφρική αλλά και στη Λατινική Αμερική, κάτι το οποίο διαπίστωσα σε πρόσφατη επίσκεψη στη Βραζιλία και στο Μεξικό. Οι ηγέτες της περιοχής των χωρών αυτών δεν είναι ηγέτες του συνόλου του πληθυσμού. Υπάρχουν περιοχές όπου εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι, αν όχι εκατομμύρια, ζουν κάτω από το κατόφλι της ε, φτώχειας και πάρα πολλές χώρες ε, είναι οι χώρες με τις μεγαλύτερες ανισότητες στον κόσμο, στη Λατινική Αμερική λέω. Και αυτά είναι διεθνή στοιχεία. Έχουμε λοιπόν ε, συμφάσεις και συμφωνίες με την περιοχή αυτή και προσπαθούμε να βοηθήσουμε κάθε χώρα για να εδρεωθεί το κράτος δικαίου και να εξαλειφθεί η φτώχεια. Δεν θα πρέπει να εγκαταλείψουμε τις χώρες αυτές. Καλό θα ήταν να επαναπροσανατολίσουμε την πολιτική συνεργασία μας. Υπ' αυτή την έννοια σας θέτω το ερώτημα, το εξή ερώτημα. Είστε υπέρ μιας ε, συνεκτικής ε, στρατηγικής ε, έτσι ώστε να έχουμε άνοδο του εισοδήματος κατά μέσο όρο στις χώρες της Λατινικής Αμερικής σε βάθος χρόνου. Σας ευχαριστώ κύριε Κορτές, λέει η Πρόεδρος. Σας λέω ότι έχετε καταχραστεί του χρόνου των υπολείπων και δεν θα έχουν την ευκαιρία να εκφραστούν. Κύριε Γκέρεντς, παρακαλώ. Πρόεδρε, μπορώ να πάρω εκείνο το λεπτάκι που δεν εξάντλησε ο Γκίμιξελ. Τις παρόλες είχε έρθει δηλαδή είχατε και... Ε, είχατε τις ευκαιρίες και άλλες φορές να αυτό μαζί, αλλά βλέπω ότι δεν το παρακάνετε κιόλα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πρώτος ε, παράγων ανάπτυξης στον κόσμο. Αριθμητική όμως είναι η δράση του, δηλαδή η συλλογή των 27 ε, κρατών μελών, των ε, παρεμβάσεων και τη συμβολή των 27 κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή των 28. Αλλά δεν αποδίδει όπως θα θέλαμε. Τα σχόλια που ακούω τώρα ε, μου αποδεικνύουν όταν φαινάκι οι ελπίδες που αισθανθήκαμε πέρυσι γιατί τώρα δεν έχουμε τα αποτελέσματα που περιμέναμε. Ενώ θα έπρεπε να είμαστε και οι πιο αποτελεσματικοί, ε, ο πιο αποτελεσματικός και ο πιο ουσιαστικός αλλά και ο πιο καθοριστικός παράγοντας ανάπτυξης στο παγκόσμιο σκηνικό καθώ είμαστε και οικονομικά ισχυρότερο. Όμω αυτά δεν τα καταφέρουμε. Πρώτον, λόγω του ρόλου του Συμβουλίου. Το Συμβούλιο έχει δύο σε υπουργικό επίπεδο συνεδριάσεις τρία ώρες το χρόνο δεν αρκούν αυτές για να μπορέσουν να ε, συγκλίνουν οι απόψεις των ε, βασικών παραγόντων που καθοδηγούν το 80% της βοήθειας για την ανάπτυξη για να γίνει αυτή η ανάπτυξη ουσία και πράξη. Δεύτερον, από τη στιγμή που αναλάβατε τα καθήκοντά σας, βλέπω να υπάρχει μια, ένα σβήσιμο θα έλεγα της φωνής του Συμβουλίου. Δηλαδή συνεδριάζει με το Συμβούλιο αλλά δεν λέει κουβέντα. Το μόνο μήνυμα το οποίο λάβαμε από το Συμβούλιο ήταν η συζήτηση για θέση εφαρμογή του άρθρου 290 της Συνθήκης Λισαβόνας. Το μόνο μήνυμα προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήταν πήγαινε δεν σαν έρχομαι. Αυτό είπε το Συμβούλιο στο Κοινοβούλιο. Δεν νομίζω ότι αυτό βοηθάει όμως ε, τον εκδημοκρατισμό, στον οποίο άλλωστε καλεί να προχωρήσουμε η συνθήκη. Και επίσης για την Επιτροπή, και το λέω και μπροστά σα, όπως και <laughs> όταν δεν είστε παρούσα, θα ήθελα για λόγους σαφήνειας και ε, αναγνωσιμότητας της κατάστασης να είναι μόνη υπεύθυνη για τον προγραμματισμό της πολιτικής ανάπτυξης η Επιτροπή γιατί χωρίς αυτό να αφαιρέσει οτιδήποτε από τι δικέ σα αρμοδιότητες, γιατί μπορείτε εσείς να περιορίσετε τον συντονισμό των πολιτικών, ενσωματώνοντας μάλιστα και ένα στοιχείο το οποίο δεν αναφέρατε στι ε, στις ομιλίες σας, ε, το εμπόριο δηλαδή. Το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί αν θέλουμε να είμαστε συνεπεί στην εξωτερική μα προσέγγιση, πρέπει και οι εμπορικέ πτυχέ να ενσωματωθούν σε αυτή την προσέγγιση. Και επίση, για τη δημοκρατία είπα ότι είχα να πω. Τελευταίο στοιχείο λοιπόν, νομίζω ότι θα πρέπει να καταβάλουμε προσπάθειες για να ικανοποιήσουμε ένα αίτημα και μια ανάγκη. Έχουμε πολύ καλές πολιτικές, ναι, θα μπορούσαν να είναι καλύτερες όμως. Εάν κάναμε τον κόπο να ε, κάνουμε το στρατηγικό σχεδιασμό πρώτα. Και αυτό είναι που λείπει, που απουσιάζει από τον ευρωπαϊκό πόλο. Καλές συζητήσεις, αλλά είναι προφανής η απουσία στρατηγικού σχεδιασμού. Και γι' αυτό σας καλώ να δώσετε στο Συμβούλιο τη δυνατότητα να ε, συμμετάσχει σε ένα διάλογο με μας για την, ε, το μελλοντικό πρόγραμμα ανάπτυξης, τη μελλοντική ατζέντα της ανάπτυξης. Είναι απαραίτητο να μιλήσουμε για τα ζωτικής αυτής και κύρια σημασία ζητήματα, γιατί ε, με το να μένει ο καθένας στη γωνιά του, στην πλευρά του, δεν πρόκειται να ενισχύσουμε την ανάπτυξη και τη στήριξη στην ανάπτυξη που ε, αναλαμβάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και Πρόεδρε, σημειώνω ότι είναι γελίο να μα περιορίσετε στα 2,5 λεπτά. Δύο φορέ το χρόνο βλέπουμε τη Λέδη Ναι, ναι, βεβαίω, μπορείτε να κάτσετε όσο θέλετε, λέει Πρόεδρο, μόνο που έχουμε ψηφοφορίε μετά. Εγώ κάθομαι και μέχρι το βράδυ, άμα θέλετε αλλά δεν νομίζω να συμφωνήσουν όλοι. Επομένως παίρνω εγώ τώρα το λόγο. θα μπορούσατε να... Δεν, δεν μπορέσατε να εκφράσετε όλε σας τις απόψεις σε τελευταία ανάλυση. Άρα δεν είστε ευχαριστημένος. Καλώς. Μου δίνω το λόγο, κυρία Άστον. Εγώ πήγα στην ΑΕΤ τρεις φορές, έξι μήνες μετά το σεισμό και μετά κατά, τη διάρκεια, κατά το δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών και τελευταία τον προηγούμενο μήνα. Δεν χρειάζεται να σας πενθυμίσω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ευρωπαίοι πολίτες επέδειξαν μια άνευ προηγουμένου ένδειξη αλληλεγγύης στο λαό της ΑΕΤΙΣ. Πλην όμως, κατά τις επισκέψεις μου αυτές και δεδομένου ότι όπως είναι γνωστό είμαστε οι κύριοι ανθρωπιστικοί χορηγοί αλλά και ανθρωπιστικοί χορηγοί για την ανάπτυξη στην ΑΕΤ ότι η συνεργασία μεταξύ ευρωπαϊκών αρχών και αρχών της, ε, της χώρας είναι πολύ περιορισμένη και αυτό το λέω με επίοικια. Μίλησα με τον Μισελ Μαρτελή, πρόεδρο τη Δημοκρατία ΑΕΤ, τον ε, Ιανουάριο στι 12 του μηνό. Συστήσαμε μεταξύ άλλων τη γεωργική πολιτική και εδώ πρέπει να πω ότι αισθάνομαι βαθύτερη ανησυχία, διότι φαίνεται ότι θέλει αυτό ο κύριο να προαγάγει μια μαζική και ε, μεγάλη έκταση γεωργία σε συνεργασία με δύο-τρει μεγάλου ομίλου, κατά πάσα πιθανότητα σε, ε, με χρήση γενετικά τροποποιημένων οργανισμών ή και υποκαταστάτων αυτών, αγνοώντα τελείω το μικρό παραγωγό και την πρόσβαση στις ΓΕΣ. Οτιδήποτε δηλαδή εμείς έχουμε προαγάγει και ε, ζητήσει από την αρχή αυτής της μεγάλης κρίσης. Θα λοιπόν τα σχόλιά σας. Ίσως να ήταν καλύτερο να απαντήσετε τώρα και μετά... Ευχαριστώ πολύ. Ε, πόση ώρα έχω για να απαντήσω. Δεν ξέρω κύριε Μίτσελ πώς μετρώνται οι επιτυχίες της αναπτυξιακής μας πολιτικής. Ο Άντρες Πίλπαλς, ο αρμόδιος επίτροπος, εξετάζει αυτά τα θέματα. Πώς μπορούμε να μετρήσουμε καλύτερα τις επιτυχίες μας. Ένα σωρό μετρήσεις μπορούμε να κάνουμε οι οποίες όμως ε, μας δίνουν ένα μέρος της εικόνας. Είναι δύσκολο να έχουμε αντικειμενικές μετρήσεις του συνόλου του συνόλου των επιτυχιών μας. Μπορούμε να έχουμε επιτεύγματα στον τομέα της εκπαίδευσης μπορούμε να έχουμε επιτυχίες διότι περισσότεροι άνθρωποι φεύγουν από την κατηγορία της απόλυτης φτώχειας και μπαίνουν στην κατηγορία π.χ. της σχετικής φτώχειας. Εν πάση περιπτώσει, γίνεται προσπάθεια να έχουμε περισσότερη συνοχή. Τα κράτη-μέλη και η Ευρωπαϊκή Ένωση στη δουλειά μας να είναι πιο συνολική. Ε, να λειτουργούμε καλύτερα. Όλα αυτά ε, είναι μέρος της ημερήσιας διάταξης που εξετάζουμε με τους ε, υπουργούς και βεβαίως ε, αξιοποιούνται τα αντίστοιχα κονδύλια. αν θέλετε θα αλλάξω τον τίτλο μου και θα γίνω foreign delegate όπως θέλετε. Ε, εν πάση περιπτώσει με τα Fiji προσπαθήσαμε να δουλέψουμε με τον τοπικό πληθυσμό για τους γνωστούς λόγους. Αν αναστείλει κανείς τη βοήθεια σε μια χώρα, τότε η περισσότερο ενδεείς είναι αυτοί που υποφέρουν και περισσότερο. Προσπαθούμε λοιπόν να έχουμε μια πιο στοχευμένη ενίσχυση και βοήθεια οι κανονισμοί για την επίγουσα κατάσταση ήταν πολύ καλοί. Τώρα όμως έχουμε ε, τους σχετικούς νόμους σε όλες τις χώρες και σε προσπαθούμε να δουλέψουμε με όλους τους οργανισμούς ούτως ώστε να ταιριάξουμε, να πλαισιώσουμε ε, καλύτερα αυτά που κάνουμε. Ως προς τη Συρία. Με την αντιπολίτευση συζήτησα διάφορα θέματα και ένα από αυτά ήταν η συμπερίληψη όλων, η εμπλοκή όλων ε, ε, όλοι όσοι προέρχονται από διαφορετικές θρησκευτικές κοινότητες και κυρίως και οι χριστιανοί θα πρέπει να νιώθουν ότι είναι μέρος της λύσης που θα βρεθεί στη Συρία και να μην νιώθουν ότι η λύση που θα βρεθεί θα αποβεί εις βάρος τους. Αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό. Το έχω συζητήσει ε, και με τους συνομιλητές μας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πώς θα διασφαλίσουμε ότι όλοι θα νιώθουν ότι έχουν συμπεριληφθεί. Ιδαλλιώς το μέλλον στη Συρία δεν θα θα, είναι μάλλον αρκετά ζωφερό. Σίγουρα στην Ιγυρία υπάρχουν πολλά παλιά θρησκευτικά ζητήματα που αναβιώνουν. Ο Goodluck Jonathan, ο πρόεδρος της χώρας αυτής, έχει εργαστεί σκληρά, προσπαθεί να βρει μια λύση. Νομίζω όμως ε, ότι πράγματι προσπαθεί να έχει μια συνολική προσέγγιση που να συμπεριλαμβάνει όλες τις ε, πληθυσμιακές ομάδες. Όλα αυτά είναι ζητήματα που ε, κρύβουν διάφορες δυσκολίες. Ένα από τα ζητήματα που συζητήσαμε με τους Υπουργούς Εξωτερικών είναι η, βεβαίως και η θρησκευτική ελευθερία και όλοι ε, δίδουν ιδιαίτερη σημασία σε αυτό. Τώρα, για τη Λιτινική Αμερική και την Κεντρική Αμερική. Ναι, πήγα εγώ στη Βραζιλία και στο Μεξικό. Αυτά τα μέρος της δουλειάς μου ως προς τις στρατηγικές εταιρικές σχέσεις και την ατζέντα για το G20. Ε, στο Μεξικό ε, συζητήσαμε την αηφόρο ανάπτυξη και τη βοήθεια ε, για την επίτευξη αυτού του στόχου. Το συζητήσαμε το θέμα αυτό και στη Βραζιλία. Σίγουρα οι χώρες αυτές έχουν πρόσβαση σε κονδύλια των αντίστοιχων ταμείων. Προσπαθούμε όμως να έχουμε μια συνεκτική στρατηγική για το σύνολο της περιφέρειας και όχι μόνο για τους στρατηγικούς μας εταίρους. Και πραγματικά καταβάλω κάθε δυνατή προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση. Από εκεί και πέρα, να σας πω και το εξής, κύριε Γκέρετς. Μετά την Λισαβόνα είναι αλήθεια ότι δεν έχουμε έρθει πολύ συχνά στην Επιτροπή σας. Ζήτησα από τον Υπουργό Ανάπτυξης της Δανίας να εμφανιστεί στην Επιτροπή σας μετά το Συμβούλιο Υπουργών Ανάπτυξης το Μάιο, αμέσως μετά, και ζήτησα και από την Κυπροϊκή Προεδρία να ε, περιλάβει αντίστοιχες προβλέψεις, γιατί ε, πράγματι θα πρέπει ε, να έχουμε στενότερη συνεργασία με την Επιτροπή για την Ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ε, ε επομένως, εάν συμφωνείτε, θα ζητήσω από τους αντίστοιχους υπουργούς να έρχονται εδώ ε, και να συζητούν μαζί σας, ελπίζοντας ότι αυτό θα αντισταθμίσει την συχνή απουσία μου από την Επιτροπή σας. Ναι. Ως αντιπρόεδρο εγώ και ο Άντρες Πίσμπαλ ως αρμόδιος επίτροπος συνεργαζόμαστε στενά, κάνουμε τα πράγματα μαζί. Ε, δεν κάνω κάτι από μόνη μου ή κάτι που να μην τον συμπεριλαμβάνει. Και εκείνο το ίδιο. Θέλουμε να έχουμε μια συνολική προσέγγιση, να έχουμε μια στρατηγική επισκόπηση αυτού που προσπαθούμε να κάνουμε. Δηλαδή, οι τη ανάπτυξη δεν εργάζονται στη γωνιά τους απομονωμένοι από όλους τους υπόλοιπους. Προσπαθούμε να προσφέρουμε ένα συνολικό πακέτο, το καλύτερο δυνατό, την καλύτερη δυνατή λύση για την κάθε χώρα. Προς αυτή την κατεύθυνση προσπαθούμε να κινηθούμε και προοδεύουμε, είναι κάτι το οποίο είναι εξελίξη. Ε, δεν είναι οριστικό και δεν έχει τελειώσει βεβαίω. Αυτή είναι η προσπάθειά μας. Τώρα για το θέμα της ITs. Τεράστια ζητήματα έχουν ανακύψει. Ε, είναι δύσκολο η κυβέρνηση να κάνει ένα βήμα προς το εμπρός. Είναι μια χώρα η οποία λαμβάνει βοήθεια τα τελευταία 50 ή 55 χρόνια και ακόμα δεν έχουν λυθεί κάποια πολύ βασικά ζητήματα. Π.χ. στις υποδομές, χτίσιμο υποδομών. Ε, προσπαθούμε να δουλέψουμε με τις τοπικές κοινότητες, να τις στηρίζουμε άμεσα να δώσουμε τη δυνατότητα στην αγροτική δραστηριότητα να αναζωπηρωθεί, ε, να αναπτυχθούν αυτές οι επιχειρήσεις και να τα συνδέσουμε όλα αυτά με την εκπαίδευση, την κατάρτιση. Τώρα, ε, το τι είδους οδιά, τι είδους καλλιέργεια θα φυτευτεί, σε τι είδου εδα, ε, δεν μπορώ να το απαντήσω τώρα. Αν θέλετε μπορώ να βρω τα στοιχεία και να επανέλθω. Ωστόσο, αυτή είναι μια χώρα η οποία αποτελεί παράδειγμα της ανάγκης ε, συνοχή στην, στην οτροπία μεταξύ κρατών μελών και Ευρωπαϊκή Ένωση και συνοχή και συνεκτική προσέγγιση μεταξύ όλων των διεθνών εταίρων. Δεν είναι θέμα απλά να χρηματοδοτούμε αυτή τη χώρα, να στέλνουμε χρήματα εκεί. Είναι να την βοηθήσουμε ουσιαστικά να ανασυγκροτηθεί ε, να χτίσει μια λειτουργική οικονομία. Και είναι βεβαίως ένα μακροπρόθεσμο εγχείρημα αυτό και θα πρέπει να δράσουμε σε όλες τις πτυχές της ε, πολιτικής ζωής. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ ο κύριος Βάγκελ έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. I have to use... Ε, δεν είμαστε πολύ αναπτυγμένοι σαν Επιτροπή, είμαι υποχρεωμένος δυστυχώς να χρησιμοποιήσω τα αγγλικά και δεν ξέρω αν θα με καταλάβετε. Δεν θα ήθελα να πάρω μέρος στην ε, περιραίουσα αρμονία. Θα ήθελα να πω ότι είχα αρκετές προσδοκίες οι οποίες μέχρι τώρα ή τουλάχιστον από την εισαγωγική της ομιλία δεν καλύφθηκαν. Θα περίμενα από πλευρά σας να αναφερθείτε σε κάποια χαίνοντα προβλήματα, σε κάποιες κρίσεις που σοβούν αυτή την εποχή και οι οποίες άμεσα επηρεάζουν αυτά τα οποία κάνουμε εδώ. Προβλήματα ανάπτυξης, προβλήματα ανθρωπιστικά, περιβαλλόμεθα στην Ευρώπη από γνωστές κρίσεις όπου υπάρχουν τα προβλήματα αυτά, υπάρχει φτώχεια, υποανάπτυξη, ανθρωπιστικές κρίσεις στην Παλαιστίνη, στον Αγκόρνο Καραμπάκ, Ξέρω ότι επαναλαμβάνομαι, αλλά εν πάση περιπτώσει θα συνεχίσω να επαναλαμβάνομαι γιατί τα προβλήματα αυτά παραμένουν. Και θα ήθελα να έρθετε κάποια φορά στη δική μας επιτροπή, στην επιτροπή ΑΦΕΤ και να μας πείτε τώρα μπορεί να νιώσετε καλά γιατί συνεισφέρομαι στο να υπάρξει η λύση ενός από όλα αυτά τα προβλήματα είτε είναι το της Δυτικής Σαχάρας, είτε είναι το Παλαιστινιακό, είτε τον Αγκόρνο Καραμπά ή κάτι άλλο. θα ήθελα να σας ζητήσω να πηγαίνετε επί τόπου να βλέπετε τα προβλήματα και το κάνετε αυτό, δεν το αποφεύγετε και αυτό είναι καλό. Πρέπει να το πούμε. Όμως θα πρέπει να προσπαθούμε και να λύνουμε τα προβλήματα, όχι μόνο να τα παρατηρούμε. και θα πρέπει όταν έχουμε ένα πρόβλημα να προσπαθούμε να μην είμαστε υποκριτές, να βρούμε τους σωστούς τρόπους για την αντιμετώπιση τους. Για τη Συρία σαν παράδειγμα και για την κριτική που ασκούμε στην τακτική του βέτο ε, των μεγάλων ε, χωρών, των ισχυρών χωρών, Κίνα και Ρωσία. Πράγματι το κάνουν αυτό οι Ρώσοι και οι Κινέζοι. Το ίδιο κάνουν και οι Αμερικανοί σε σχέση με τα δικά τους συμφέροντα και δεν διαμαρτυρόμαστε γι' αυτό, τους βοηθάμε. Λοιπόν, δεν θα πρέπει να κάνουμε κριτική στους άλλους για κάτι που κάνουμε και εμείς οι ίδιοι. Ελπίζω να με καταλάβατε και ελπίζω να έρχεστε στο μέλλον με συγκεκριμένες πρωτοβουλίες για το πώς θα λύνονται κάποια από τα προβλήματά μας. Κέλλερ. Ευχαριστώ μετά από αυτή την εισαγωγή στον κόσμο θα ήθελα να επιστρέψω στις ευρωπαϊκές πολιτικές. Έχω πολλές ερωτήσεις, θα προσπαθήσω όμως να είμαι σύντομη. Πρώτον, θα ήθελα να μάθω πώς ακριβώς αντιμετωπίζετε με το θέμα των πιστώσεων για την ανάπτυξη. Πώς ακριβώς προχωράτε στο mainstreaming των πολιτικών σας τι κάνετε με το μνημόνιο συνεργασίας ανάμεσα στη Γενική Διεύθυνση ΔΕΦΚΟ και στην υπηρεσία σας εξωτερικής δράσης. Αναφερθήκατε στο πόσο πολύτιμο είναι να υπάρχει συνεισφορά και από πλευρά του Κοινοβουλίου και η αλήθεια είναι ότι μερικές φορές πράγματι είμαστε χρήσιμοι. Ποτέ όμως δεν το λαμβάνετε υπόψη. Όταν κοιτάμε τα προγράμματα, τα έγγραφα για τη στρατηγική, στρατηγικά συγγνώμη, έγγραφα για διάφορες χώρες δεν βλέπουμε τη δική μας συνεισφορά πουθενά. Θέλουμε να έχουμε πρακτικές δυνατότητες για να επηρεάσουμε την κατάσταση είτε μέσω των κατεξουσιοδότηση πράκτεων, πράξεων είτε με άλλο τρόπο. Πρέπει να προσπαθήσουμε δηλαδή να σας στηρίξουμε, αλλά πρέπει να βρούμε και τους τυπικούς τρόπους για να το κάνουμε. Τέλος, υπάρχει λοιπόν μπροστά μας μια ατζέντα για αλλαγή και ο κύριος Πίμπαλξ έχει προωθήσει την ατζέντα αυτή. Μας είπε ότι δεν αντικαθιστά τη συνένεση που υπάρχει την πολιτική για την ανάπτυξη, αλλά ένας εκπρόσωπος της Επιτροπής σήμερα το πρωί είπε η νέα μας πολιτική στην ανάπτυξη είναι η ατζέντα για την αλλαγή. Εδώ φαίνεται κάτι καινούριο μπροστά μας. Ίσως η συνένεση στην οποία είχαμε καταλήξει να μην είναι τόσο έγκυρη ή έγκριτη όπως το παρελθόν. Τι θέση έχετε λοιπόν σε σχέση με την ατζέντα για αλλαγή από δική σας σκοπιά. Πώς το βλέπετε. Έχετε ξεκινήσει την εφαρμογή αυτών που προβλέπονται στα πλαίσια αυτής της ατζέντα για αλλαγή της νέας πολιτικής. Αναφέρεται σε θέματα διακυβέρνησης. Δεν είναι κάτι το πλήρες σε αυτή τη φάση. Αλλά μήπως υπάρχουν κάποιες αντιφάσεις εδώ σε σχέση με αυτό που ονομάζουμε το ποιοι είναι υπεύθυνοι για την ανάπτυξη, ποιοι είναι σε εισαγωγικά ιδιοκτήτες για την ανάπτυξη. Πολλές ερωτήσεις, συγγνώμη. Ντίβα, ευχαριστώ Πρόεδρε. Σας συγχαίρω, κάνατε ό,τι μπορείτε αυτή την περίοδο και για το Σουντάν, μπορέσατε και περιορίσατε τον πρόεδρο Μπασίρ. Ξέρετε ότι είναι υπεύθυνο για τη δολοφονία καθημερινά, ακόμα και σήμερα ανθρώπων από ό,τι συμβαίνει στη Συρία αλλά οι εφημερίδες δεν ασχολούνται με το Σουδάν. Εσείς όμως ασχολείστε με το Σουδάν και σας είμαι ευγνώμων. Λοιπόν, θα πάω γρήγορα. Τρεις ερωτήσεις. Πρώτον, για τα θέματα της διαφθοράς. Η Επιτροπή μας έχει πει ότι 700 δις δολάρια μαύρο χρήμα εισάγεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις δυτικές οικονομίες από τις αναπτυσσόμενες χώρες κρυφά βρώμικα, ματωμένα λεφτά οι Ινδοί από ό,τι φαίνεται από μόνο έχουν δύο-τρει ε, ε, σε ελβετικού λογαριασμούς. 700, εκατομμύρια, 700 δις ευρώ μιλάμε για δύο φορές τον κοινοτικό προϋπολογισμό. Δίνουμε σε αυτές τις χώρες 60-70 δις και παίρνουμε από τις χώρες αυτές σε μαύρο χρήμα αφορολόγητο 10 φορές το ίδιο ή 7 φορές το ίδιο. 7 φορές διορθώνει ο μιλητής το ίδιο. Τι μπορούμε να κάνουμε λοιπόν, μήπως τα χρήματα αυτά θα μπορούσαν να είναι πιο χρήματα, πιο χρήσιμα στις περιοχές αυτές τώρα. Αργεντινή. Σήμερα διαβάσαμε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο δίδει στην Αργεντινή 450 εκατομμύρια βοήθεια λίρες. Και ταυτόχρονα οι Αργεντινοί μας απειλούν και απειλούν το Ηνωμένο Βασίλειο για το θέμα των Φόκλαντς. Ε, πώς μπορούμε να δίνουμε λεφτά στους Αργεντίνους για βοήθεια την οποία μπορεί να χρησιμοποιήσουν για να εξοπλιστούν και να επιτεθούν στα νήσους Φόρκλαντς. Αυτό είναι απαράδεκτο. Μια τελευταία ερώτηση για τις ε, λίμνες υψηλού υψομέτρου στα Χιμαλάια, τις αλπιτής ε, λίμνες που σχηματίζονται από από τους παγετώνες. Έχουν δημιουργηθεί κάποιες νέες τέτοιες λίμνες από την τήξη των παγετώνων και 200 εκατομμύρια κόσμος απειλείται και στην Ινδία και στην Κίνα. Τι θα κάνετε γι' αυτό. Ευχαριστώ κύριε Ντίβα, ο κύριος Κατσμαρέκ. Ευχαριστώ για την παρουσία σας Αντιπρόεδρε. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω επίσης και για την απόφαση η οποία ελήφθη χθε για τη Λευκορωσία και την ανάκληση των πρέσβεων από το Μίνσκ. Το θέμα αυτό ε, δεν συνδέεται τυπικά μόνο με την αναπτυξιακή βοήθεια. Η απόφαση που ελήφθη ήταν μονομερής και κατάλληλη σε σχέση με την κατάσταση. Και νομίζω ότι είναι συμβατό με τους στόχους της δημιουργίας της υπηρεσίας εξωτερικής δράσης, έτσι ώστε να παίρνει γρήγορες και κατάλληλες αποφάσεις. Στην περίπτωσή μας, στην περίπτωση της Λευκορωσίας ήταν πολύ καλή η δράση αυτή, μονομερής μεν, αλλά κατάλληλη και γρήγορη. Τώρα, μια ερώτηση για το μέλλον. Όπως γνωρίζετε, κυρία Άστον, έχει πολύ μεγάλη σημασία για τους στόχους της, ανάπτυξης, της συνεργασίας για τις ανάπτυξης είναι οι στόχοι της χιλιετίας. Οι στόχοι της χιλιετίας πρέπει να ολοκληρωθούν μέχρι το 2015. Παρ' όλα αυτά οι διαπραγματεύσεις σε επίπεδο ΟΗΕ έχουν ξεκινήσει για το τι θα γίνει μετά το 2015. Πρόκειται για ένα στρατηγικό θέμα θα έλεγα τι θα γίνει ε, με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ποιος θα είναι ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά το 2015 και πώς θα συνεχίσουμε να συνεισφέρουμε στους στόχους της χιλιετίας μετά το 2015. Η Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πράγματι υπάρχουν πολλά προβλήματα και λέτε πρέπει να έλθω εδώ με λύσεις. Θα πρέπει να αναγνωρίσουμε δύο, δύο θέματα εδώ. Πρώτον, η Ευρωπαϊκή Ένωση παίζει ένα πολύ ουσιαστικό ρόλο και στο Παλαιστινιακό, στα πλαίσια μάλλον της προσπάθειας της Παλαιστινιακής Αρχής να οικοδομήσει τους θεσμούς του νέου κράτους, και στηρίζουμε επίσης και τις προσπάθειες συνεννόησης ανάμεσα στο Ισραήλ και την Παλαιστίνη που θα οδηγήσει στη λύση των λεγόμενη λύση των δύο κρατών. Το δεύτερο θέμα που θέσατε είναι τον Αγκόρνο Καραμπάχ. Είχα πάει πρόσφατα στο Αζερβαϊτζάν και την Αρμενία για να προσπαθήσουμε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε έτσι ώστε να υπάρξει περισσότερη εμπιστοσύνη ανάμεσα σε αυτές τις χώρες γιατί υπάρχουν πολλά προβλήματα στη συνοριακή τους γραμμή. Είναι κάτι το οποίο με ανησυχεί ιδιαίτερα αλλά οι λύσει θα πρέπει να γίνουν αντικείμενο συμφωνίας ανάμεσα στα άμεσα εμπλεκόμενα μέρη. Εγώ έκανα ορισμένε προτάσει και για του Παλαιστινίου και του Ισραηλινούς, δεν μπορώ να του υποχρεώσω να συμφωνήσουν βέβαια. Αυτό το οποίο μπορούμε να κάνουμε όμως είναι να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε σκληρά και με τους Ισραηλινούς και τους Παλαιστινίους και τους Ιορδανούς και με τους Αρμένιους και ε, τους κατοίκους του Ναγκόρνο Καραμπάχ από την άλλη έτσι ώστε να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε μια λύση την οποία να στηρίξουμε όλοι. Αν είχα ένα μαγικό ραβδί το οποίο θα κινούσα θα το έκανα αυτό. Έχω πάει στην περιοχή αυτή τρεις φορές τον τελευταίο καιρό, θα συνεχίσω και περιμένετε να συνεχίσω να πηγαίνω και θα το κάνω. Βλέπουμε ποια είναι η τραγική πλευρά αυτού του είδους των συγκρούσεων Παρ' όλα αυτά πετύχαμε αρκετά πράγματα, πράγματα τα οποία δεν είναι αρκετά από μόνα τους, αλλά τα οποία βοηθούν να αλλάξουν προς το καλύτερο τα πράγματα. Δεν παρετούμεθα. Αλλά δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις. Δεν μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση με μαγικά τρίκ να λύσει τα προβλήματα. Αυτό το οποίο μπορεί να κάνει είναι να υπογραμμίσει την επιμονή μας στον σεβασμό του διεθνούς νόμου. Πιστεύουμε ότι οι λαοί της Αρμενίας και του Αζερβαϊτζάν πρέπει να βρουν μια λύση και ακριβώς η προσπάθειά μας είναι να τις βοηθήσουμε τις χώρες αυτές να καταλήξουν σε μια συμφωνία. Έχουμε ένα ειδικό εκπρόσωπο με τις δύο αυτές χώρες και με τη Γεωργία, αλλά λύση μαγική δεν υπάρχει. Το ίδιο ισχύει και για τη Δυτική Σαχάρα. Εμείς στηρίζουμε τις διαδικασίες των Ηνωμένων Εθνών. Μερικές φορές ε, η σύραξη αυτή φαίνεται ή φέρεται ότι είναι μια παγωμένη σύραξη, αλλά δεν το πιστεύω, εμένα μου φαίνεται ότι διόλου παγωμένη δεν είναι. Το θέμα είναι να βρούμε μια λύση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση όμως αναγνωρίζεται στις περιοχές αυτές για αυτό το οποίο κάνει και στο Μεσανατολικό και αυτό γίνεται χάρη και στις δικές σας προσπάθειες. Αλλά τις λύσεις θα τις βρουν οι άμεσα εμπλεκόμενοι. Και πιέζουμε προς την κατεύθυνση αυτή κυρία Κέλλερ. Θέσατε πάρα πολλά θέματα, ίσως δώσω κάποιες απαντήσεις. Όταν άρχισα να ακούω τα θέματα της συνεκτικότητας της πολιτικής μας δράσης στην ανάπτυξη, χρειάστηκα χρόνο. Χρειάστηκα χρόνο γιατί απαιτείται να υπάρξει συνεκτικότητα των πολιτικών μας. Εμπόριο, επενδύσεις, κλιματολογικές αλλαγές, το πώς προσπαθούμε να δράσουμε στα πλαίσια όλων αυτών των πολιτικών εξελίξεων που έχουν σαν την ανάπτυξη. Η ανάπτυξη όμως δεν είναι μόνο βοήθεια. Η ανάπτυξη είναι όλα τα πράγματα τα οποία μπορούν να δημιουργήσουν νέες διαφορετικές καταστάσεις. Σε αυτό αναφερόμουν. Πώς μπορεί κανείς να τα συνδυάσει όλα αυτά. Πώς μπορεί να έχει στρατηγική ανάπτυξη, αναπτυξιακή τέτοια έτσι ώστε οι χώρες ε, να πετύχουν τις οποίες θέλουμε να βοηθήσουμε στους στόχους τους και δημιουργώντας και οικοδομώντας δημοκρατικούς θεσμούς, αποκαθιστώντας το κράτος δικαίου, την κοινωνία των πολιτών, όλα αυτά τα οποία μπορούν να ε, βοηθήσουν τις χώρες ε, και στον τομέα των σχολείων και στον τομέα ε, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων κτλ. Εμείς και η Επιτροπή προσπαθούμε να βοηθήσουμε προς την κατεύθυνση αυτή. Δεν είναι τέλεια τα πράγματα βέβαια, αυτά τα οποία κάνουμε, αλλά είναι ό,τι καλύτερο σε αυτή τη φάση μπορούμε. Έχουμε σωστές μορφές συνεργασίας με το EIS. Δεν έχω ακούσει να υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα, αλλά όπως είπα στην αρχή, αυτό το οποίο μπορούμε να κάνουμε εν μέρη τουλάχιστον είναι να βρούμε νέους τρόπους, νέες υπηρεσίες. Δεν νομίζω ότι αυτά τα οποία προτείνεται δεν λαμβάνονται υπόψη από αυτά τα οποία κάνουμε εμείς επανειλημμένα από ό,τι εγώ γνωρίζω, ακούω για ιδέες, ακούω για προτάσεις, ακούω για αποφάσεις οι οποίες προέρχονται από εσά, έχουν ξεκινήσει από εσά, από το Κοινοβούλιο. Αυτό το οποίο δεν κάνουμε ίσως είναι να επικοινωνούμε τόσο συχνά όσο έπρεπε. Τώρα για τις κατεξουσιοδότηση πράξεις τις υποστηρίζω. Εγώ δεν ε, λαμβάνω τις αποφάσεις για αυτές τις πράξεις, αλλά παρόλα αυτά θεωρώ ότι διευκολύνουν την εμπλοκή με την οποία εμείς ε, μπορούμε να έχουμε στα πλαίσια των δημοκρατικών θεσμών. Τώρα για την ατζέντα για αλλαγή. Είπατε αν αντικαθιστά την πολιτική συνένεση η οποία υπάρχει. Όχι, τη συμπληρώνει. Θέλουμε τα πράγματα να δουλέψουν καλύτερα, θέλουμε τα πράγματα να πάνε καλύτερα, θέλουμε να βρούμε τρόπους έτσι ώστε να χρησιμοποιήσουμε τους όρους, τους πόρους τους οποίους έχουμε με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο. Και έρχομαι σε αυτά τα οποία έλεγα πριν. Πώς μπορεί κανείς να υπολογίσει αυτά τα οποία γίνονται, πώς μπορεί να πιστέψει ότι αυτά τα οποία διαθέτει για βοήθεια χρησιμοποιούνται σωστά. Όταν βοηθάς τους ανθρώπους στην βάση, καλύπτεις τις προσδοκίες τους, αλλά πρέπει να είσαι σίγουρος για την επιτυχία των προσπαθειών σου. Για τον κύριο Ντίβα το να μένουν τα χρήματα σε αυτές τις χώρες. Το θέμα είναι πολύ ενδιαφέρον, γιατί από τη μία το να βοηθά κανείς τις χώρες αυτές μέσω του προϋπολογισμού είναι στην ουσία έχει σαν στόχο να βοηθήσουμε τις χώρες να δουλέψουν από μόνες τους, να λειτουργήσουν από μόνες τους. Έχουμε κάνει ενδιαφέρουσες συζητήσεις με το ελεγκτικό συνέδριο για αυτά τα θέματα. Πρώτον αυτό που μπορούμε να κάνουμε και το οποίο εγγράφεται στα πλαίσια της νέας στρατηγικής ας πούμε γειτονίας είναι τα χρήματά μας να πηγαίνουν εκεί που πρέπει. Οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών θέλουν να υπάρχει μια βεβαιότητα σε σχέση με το πού πηγαίνουν τα χρήματα και ποιοι είναι υπόλογοι για τον τρόπο με τον οποίο θα δαπανηθούν τα χρήματα αυτά. Πρέπει να προσπαθήσουμε λοιπόν να προωθήσουμε τις σχέσεις μας με τις χώρες εταίρους με αποτελεσματικό τρόπο έτσι ώστε τα χρήματα που διαθέτουμε να φτάνουν εκεί που πρέπει. Υπάρχουν και ευρύτερα θέματα που τίθενται από τις ερωτήσεις σας, τις οποίες, τα οποία θέματα δεν μπορώ εγώ ίσως να σχολιάσω και να απαντήσω. Αν φάρω το παράδειγμα της Ομαλίας, βλέποντας από πού προέρχονται τα χρήματα, έχει σημασία το να παρακολουθήσει κανείς την τροχιά των χρημάτων αυτών. Ιδιαίτερα τα χρήματα τα οποία έχουν σαν στόχο την καταπολέμηση της πειρατείας για την Αργεντινή. Όπως ξέρετε το θέμα αυτό είναι ένα διμερές θέμα ανάμεσα σε δύο κυρίαρχα κράτη. Αυτό το οποίο θα πω είναι ότι υπάρχουν άνθρωποι και στην Αργεντινή όπως και σε όλες τις χώρες που βοηθάμε τους οποίους προσπαθούμε να καλύψουμε τις ανάγκες τους στον τομέα της εκπαίδευσης κτλ. Και αυτό είναι για μένα το οποίο πρέπει να λάβουμε υπόψη μας, ανεξαρτήτως αυτών που συμβαίνουν σε επίπεδο πολιτικό. Τώρα για τις λίμνες από τους παγετώνες που λιώνουν στα Ιμαλάια δεν ξέρω να σας δώσω, δεν έχω να σας δώσω απαντήσεις. Κοιτάξτε, εμείς προσπαθούμε να ομαδοποιήσουμε κάποιες χώρες να αντιμετωπίσουν θέματα που τις επηρεάζουν άμεσα. Υδάτινοι πόροι, κλιματολογικές αλλαγές, όλα αυτά είναι θέματα τα οποία άπτονται και της ενέργειας και προσπαθεί κανείς να φέρει σε επαφή τις χώρες έτσι ώστε να τα αντιμετωπίσουν, των περιοχών αυτών για να τα αντιμετωπίσουν. Για τον κύριο Κάτσμαρεκ, Λευκορωσία. Πράγματι, η απόφαση ελήφθη πάρα πολύ γρήγορα, δεν ήταν δύσκολο να ληφθεί η απόφαση αυτή. Μερικέ φορέ οι αποφάσει απαιτούν περισσότερο χρόνο γιατί είναι πιο δύσκολε. Τώρα όχι. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι εμεί θα συνεχίσουμε να βοηθάμε τον λαό τη Λευκορωσίας, να πιέζουμε για την απελευθέρωση των φυλακισμένων Λευκορώσων. Εμεί ε, το ξεκαθαρίσαμε αυτό στον πρόεδρο τη χώρα, όταν ο πρέσβη μα προσεκλήθη να επιστρέψει μαζί με τον Πολωνό πρέσβη Όλες οι χώρες θεώρησαν ότι θα κάνουν το ίδιο και θα αποσύρουν και αυτοί τις, ε, τους πρέσβες τους. Νομίζω είναι ένα καλό παράδειγμα συνεργασίας. Τώρα για τους στόχους της χιλιετίας. Πολλά έχουν αρχίσει να γίνονται τώρα σε σχέση με το μέλλον. Έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία να έχουμε τους σωστούς στόχους και να δούμε πόσο μπορούμε να προχωρήσουμε προς την κατεύθυνση αυτή. Σαν παράδειγμα, στον τομέα... Στο um, I hope της υγείας ε, των γυναικών, των μητέρων, προσπαθούμε τα χρήματα αυτά να βοηθήσουν. Θα τα συζητήσουμε τα θέματα αυτά στη συζήτηση για το νέο πλαίσιο. Σας ευχαριστώ, κύριος Μαρτίνες. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω και την Κάθη και να κάνω τα εξής σχόλια και να θέσω τις ε, εξής τρεις ερωτήσεις. Ποια είναι η άποψή σου, Κάθη, για την κοινοβουλευτική διάσταση των πρεσβειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των αντιπροσωπιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή, αντί για αντιπροσωπείες της Επιτροπής, έχουμε ουσιαστικά πρεσβείες ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι μόνο της Επιτροπής. Άρα, ενδεχομένως, ε, θα πρέπει και οι αντιπροσωπείες ε, σε κάθε σημείο εκπροσώπησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανά τον κόσμο να μπορούν να είναι υπόλογες και στο δικό μας κοινοβούλιο. Και ενδεχομένω θα πρέπει κάποιοι άνθρωποι να ασχολούνται με τα κοινοβουλευτικά θέματα που έχουν να κάνουν τη συγκεκριμένη χώρα και να μπορούν να χαίρουν τη δική μα στήριξη. Είναι λίγο παράδοξο αυτό, αλλά έχω να πω το εξή. Εκεί όπου η πρέσβη είναι διπλωματική, στελέχη του διπλωματικού σώματος, ε, πάντοτε ε, διάκειται ευμενώς έναντι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ενώ όταν είναι πρώην στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, αμελούν θα έλεγα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτό καταρχάς. Κατά δεύτερο, μία πολύ ενδιαφέρουσα περιφερειακή διάσκεψη έγινε με τις χώρες ΑΚΕ και την Νότια Αφρική και τα λοιπά, πολύ πρόσφατα. Και τέθηκαν θέματα πολύ σημαντικά συζητήσαμε με τους πρέσβεις από όλα τα κράτη-μέλη και τους ρώτησα το εξής. Πιστεύετε ότι από τη συνθήκη της Λισαβόνας και μετά λειτουργείτε καλύτερα ως ομάδα. Και μου απάντησαν ναι, λειτουργούμε καλύτερα ως ομάδα, αλλά ε, δεν το έχει αυτό υπόψη της η κοινή γνώμη και οι αρχές ε, στη Ζάμπια. Δηλαδή, δεν έχουν την αντίληψη ότι ε, λειτουργεί συντονιστικά η Ευρωπαϊκή Ένωση και ότι δεν έχουν να κάνουν με κάθε μια χώρα ξεχωριστά, Γαλλία, Γερμανία κλπ. Και άλλα πράγματα είδαμε, ότι διεξάγονται τρεις αγώνες πολύ σημαντικοί στην Αφρική. Η πρώτη μάχη είναι η απόκτηση περισσότερων δυνατοτήτων ε, από τις γυναίκες, το empowerment που λέμε. Αυτή τη μάχη την κερδίζουμε. Οι γυναίκες προχωρούν, είναι η παρουσία τους όλο και πιο στεναρή. Είναι μια μάχη που κερδίζουμε καθημερινά και αυτό είναι πολύ θετικό. Δεύτερη είναι η μάχη ενάντια στο AIDS. Έχουμε σημειώσει πρόοδο, αλλά αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε τέλμα. Και τρίτη μάχη είναι μια μάχη που με απασχολεί ιδιαιτέρως, η μάχη ενάντια ε, στην ομοφοβία. Δηλαδή, επέστρεψα από τη Λουσάκα και πραγματικά... Ε, Ήρθε ο κύριος Μπανκιμούν, απευθύνθηκε στο κοινοβούλιο και είδα την αντίληψη της κοινή γνώμης και την αντίληψη των εκπροσώπων ε, των εθνικών αρχών ασκεί το πολύ μεγάλη ε, κριτική στον παρκιμούν, πριν καν να, να πάρει το λόγο για το ενδεχόμενο ε, να αναφερθεί στα δικαιώματα των ομοφιλοφιλών και το καθεξής. Και στο τέλος να πω ότι έχετε δίκιο ότι ε, Έχετε δίκιο ότι μιλάτε πολύ καλά αγγλικά, αλλά δεν είναι το θέμα πόσο καλά αγγλικά μιλάει κανείς, αλλά τι ακριβώς λέει στα αγγλικά. Ευχαριστώ πολύ, Κάθη, η Πρόεδρος. Ευχαριστούμε. Κύριε Σας ευχαριστώ που αποφασίσατε να επανέλθετε εδώ. Η συμμετοχή σας για μας είναι πολύ σημαντική. Είναι κάτι το οποίο όλοι θέλουμε και γι' αυτό θέλουμε να σας βλέπουμε και πιο συχνά. Έχω προετοιμάσει ένα ερώτημα για την Αιτία, αλλά τέθηκε από την πρόεδρό μας και σας ευχαριστώ για την απάντηση. Πράγματι δεν έχω κάτι άλλο να πω, κερδίσατε τουλάχιστον δύο λεπτά. Ευχαριστώ κυρία Ζανίκη. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Νιούτον Τάν. Κι εγώ πολύ σύντομα πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε και πάλι επαναλαμβάνω την ε, πρόταση να μας ξαναεπισκεφθείτε. Δεν είσαστε συνήθως στις Βρυξέλλες, συνήθως κυκλοφορείτε ανά τον κόσμο, αλλά πάντως ευχαριστούμε που είστε εδώ. Ε, μαζί με άλλου δύο συναδέλφου, των οποίων ένα είναι εδώ σήμερα, πήγαμε στην Ινδία για να επανεξετάσουμε την ανάγκη για, να, ε, για περαιτέρω βοήθεια ή ο συντονισμό τη βοήθεια προ την Ινδία. Και ο Ικανό και ο στη δική του ανάλυση. Καταλαβαίνω αυτό που λέτε, ότι είναι πολλέ οι περιπτώσει όπου σε ορισμένε χώρε ε, ο κόσμο δεν παίρνει τη βοήθεια που αποστέλλεται, όπω παραδείγματι στην Ινδία. Από 500 εκατομμύρια, είναι οι Ινδοί, οι με κάτω από ε, μισό ευρώ την ημέρα. Μην ξεχνάμε ότι όταν ε, αναπτύσσονται έργα, αυτά πολύ συχνά τα έχει χρηματοδοτήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μεν, πλην όμω ο κόσμο δεν έχει καν ιδέα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Άρα λοιπόν, όταν το ΕΚΟ χρηματοδοτεί χρήματα, καλό θα είναι να λέει Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι Κομισιόν, Κοινοβούλια, Υπηρεσία Εξωτερική Δράση. Ένα απλό αίτημα, να καταλαβαίνει ο κόσμο σε τι πράγμα αναφέρεται. Καλώς λέει η Πρόεδρος, η κυρία Τσίμερ. Σας ευχαριστώ. Ως μέλος της Επιτροπής, έχω συλλέξει την εμπειρία ότι οι προσδοκίες ε, ότι η πολιτική για την ανάπτυξη θα είναι συνεπής μαζί με άλλες πολιτικές ε, διαψεύεται διαρκώς τελικά διαπιστώνουμε ότι στους διάφορους τομείς αναπτύσσονται συμφέροντα εθνικά, ακόμα δε και με απεικιοκρατικό χρωματισμό συμφέροντα και στην αναπτυξιακή πολιτική και σε άλλες. Τώρα λοιπόν έχουμε το τρίγωνο πολιτική ασφάλειας, εμπορική πολιτική, πολιτική για την ανάπτυξη. Η αναπτυξιακή πολιτική σε αυτό το μαγικό τρίγωνο φαίνεται να χάνεται, σαν να την έχει απορροφήσει το τρίγωνο των Βερμούδων. Η εμπορική πολιτική φαίνεται από την άλλη να παίρνει το πάνω χέρι και η αναπτυξιακή μας πολιτική μετατρέπεται σε μια πολιτική αναπτυξιακή με γνώμονα μόνο το εμπόριο. Δηλαδή μετατρέπεται σε ένα μέσον για να διασφαλίζονται πόροι και πρόσβαση στις αγορές. Αυτή είναι η εντύπωσή μου. Και γι' αυτό σας ερωτώ το εξή. Πώς αξιολογείτε τον ε, περιορισμό ιδιαίτερα στο ζήτημα της ε, πρόσβασης στις αγορές για τις ε, λιγότερο ανεπτυχημένες χώρες, LTC. Τι σημαίνει αυτό, η περιορισμένη πρόσβαση αγορές. Έχετε επαληθεύσει συνέπειες, έχετε μπορέσει να δείτε αν υπάρχει προσμετρήσιμη ε, αξία της ανάπτυξης Έχετε συγκεκριμένα κριτήρια για το πώς μπορεί η κατάσταση προς την ανάπτυξη να καταμετρηθεί, να ποσοστοποιηθεί, όπως και σε αντιπαράθεση με τις upper income countries, τις χώρες δηλαδή του υψηλότερου επίπεδου και βεβαίως ε, σε συσχετισμό με είτε φυσικές καταστροφές είτε εμπόλεμες καταστάσεις οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν σημαντικά το εισόδημα των κρατών αυτών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Η αντιπροσωπεία είναι στη θέση σα, κύριε Μαρτίνε, όπω και κάθε αντιπροσωπεία τη Ευρωπαϊκή Ένωση, ανά τον κόσμο, είναι στην υπηρεσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σε κάθε αντιπροσωπεία υπάρχει κάποιος υπάλληλος υπεύθυνο για τις επαφές με το Κοινοβούλιο, contact point και με χαρά πάντοτε λαμβάνω μηνύματα βουλευτών όταν ε, μου λένε ότι ήταν ικανοποιημένοι από την υπηρεσία, από την εξυπηρέτηση των, ε, του προσωπικού αυτού και πάνω απ' όλα θέλω να βλέπω τα μηνύματα αν τυχόν δεν ήσασταν ικανοποιημένοι. Για τη διάσκεψη των επικεφαλής των αντιπροσωπιών και τις συνομιλίες ε, με αυτούς πρέπει να επισημάνω ότι αυτό αποτελεί κομμάτι της δουλειάς. Δηλαδή ε, πρέπει να βεβαιωνόμαστε πάντοτε ότι πρέπει ε, να ε, ότι διαρκώς αναπτύσσεται η υπηρεσία μας και προσπαθώ πάντοτε να ενισχύω και τους δεσμούς μεταξύ των μελών του προσωπικού μας, ελπίζοντας ταυτόχρονα ότι η συνεργασία στην πράξη ανά τον κόσμο λειτουργεί ικανοποιητικά Πάντα βέβαια περιμένω και τα δικά σας σχόλια, καθώς η δική μου πόρη επαλήθευσης είναι περιορισμένη. Για την συνεδρίαση ΑΚΕ στην Ουσάκα, στην Ουσάκα. Ε, προσπαθούμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση να κερδίζουμε από τη συνεργασία, την ομαδική συνεργασία Ευρωπαϊκή Ένωση και κρατών, Ευρωπαϊκής Ένωσης και κρατών μελών. Πρέπει να είναι σαφές δηλαδή ότι είμαστε μία ομάδα, δεν ανάγκη να μένουμε σιωπηλοί είτε ο μεν είτε ο δε. Αλλά να λέμε πάντα το ίδιο πράγμα όταν λέμε κάτι. Ε, Μεξικό Φερρυπίν, όπου ξέρετε, εγώ συναντώ και όλους τους πρεσβευτές από, τους, ε, από τα κράτη-μέλη που εκπροσωπούνται υπό την Προεδρία της Αντιπροσωπείας ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο Μεξικό λοιπόν το μήνυμα και επαναλαμβάνεται σε όλες τις χώρες του κόσμου είναι πόσο καλή ήταν η δουλειά, ο συντονισμός ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι όλο και πιο ισχυρό το μήνυμα αυτό. Διότι πολλέ φορέ όλοι κάνουν την ίδια κίνηση σαν ε, μία ομάδα. Και αυτό βέβαια ακόμα και ότι το, το να μπαίνει κανεί μέσα στην αίθουσα ομαδικά είναι, σαν, ε, είναι πάρα πολύ εντυπωσιακή κίνηση. Έχουμε 14 μήνε ε, δουλειά στην υπηρεσία αυτή. Σε 5-10 χρόνια διανοηθείτε τι προόδου μπορούμε να σημειώσουμε, τι μεγάλο αντίκτυπο μπορούμε να εξασφαλίσουμε και πόσο καλύτερα μπορούν να δουλεύουν οι υπηρεσίε μα στι διάφορε χώρε. Πάντω εγώ σε κάθε μου επίσκεψη ε, ξετάζω και επαληθεύω πώς είναι η δουλειά μας στην χώρα αυτή, πώς βλέπουν οι αντιπροσωπ... τις αντιπροσωπείες μας οι κυβερνήσεις και το καθεξής. Για το θέμα της ε, απόρριψης ή του φόβου των ομοφιλοφίλων ε, των ε, λεσβιών, γενετικά ε, παρενδυτικών και άλλων. Ξέρετε ότι ε, είναι ένα θέμα το οποίο με ενδιαφέρει ιδιαίτερο. Το έχω προαγάγει και νομοθετικά και είμαι, πρέπει να πω ότι είμαι υπερήφανη που ήμουνα από τους πρώτους ή πρώτοι πολιτικός που το προώθησε το ζήτημα αυτό στα δρομία μου. Είναι ένα θέμα λοιπόν το οποίο πρέπει σε κάθε περίπτωση για διάφορους λόγους, είτε πρόκειται για προκαταλήψεις ιστορικές, ιστορικούς λόγους, ε, πολιτιστικούς ή άλλους, να αντιμετωπίσουμε όπου υπάρχουν ακόμα προβλήματα, υπάρχει ανάγκη για να αντιμετωπίσει το θέμα αυτό. Και φαντάζομαι ότι στην Λουσάκα και ο Μπαν Κιμούν αυτό προσπαθούσαν να κάνει, να συστήσει ακριβώ αυτό το θέμα. Η δική μου θέση είναι ξεκάθαρη και δεν έχω σιωπήσει ποτέ στην υπόθεση αυτή. Ο Νιούτον Ντάν και η Ινδία, καθώ η κυρία Ζανουσίου έχει αποχωρήσει. Υπάρχει πολλή δουλειά που γίνεται στην Ινδία. Για διάφορου λόγου. Πρώτον, έχουμε αρκετή δουλειά ω προ την υποστήριξη. Και υποστήριξη, από την άλλη, δεύτερον, προ την κυβέρνηση ώστε αυτή με τη σειρά τη να κάνει το μερίδιο της δουλειά ε, που τη ανήκει για την ανάπτυξη. Ναι. Ε, δεν συμφωνώ ότι το εμπόριο επικρατεί σε σχέση με την ανάπτυξη, αλλά θα το συζητήσουμε. η εικόνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το αν θα λέμε Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή κάτι άλλο. Προφανώς αυτό είναι ένα παλιό πάνω, μια παλιά πινακίδα και δεν μπορούμε να διανοηθούμε ότι θα αλλάξουμε κάθε πινακίδα ανά τον κόσμο. Αλλά από εδώ και προς τα καινούργια έργα πάντα λένε Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν έχει σημασία κανείς να γνωρίζει αν είναι Συμβούλιο, Κοινοβούλιο ή Επιτροπή, αρκεί να ξέρει ότι είναι Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης ε, για το ποιος καθοδηγεί την ανάπτυξη το εμπόριο, το περιβάλλον. Δεν συμφωνώ με τη δική σας ανάπτυξη γιατί δεν θεωρώ ότι μπορεί να υποβιβαστεί η σημασία του να βοηθήσουμε τις χώρες αυτές στην ανάπτυξη των δικών τους, ε, του δικού τους δυναμικού, δηλαδή να αναπτύξουν οικονομία αυτόνομη, με εμπορικές σχέσεις αυτόνομες. Εάν είστε στην Αφρική τη μεγάλη σημασία της ανάπτυξης ενδοαφρικανικών εμπορικών σχέσεων, πόσο σημαντικό μπορεί να είναι για την ανάπτυξη των οικονομιών αυτών, των λαών αυτών. Και αυτό το λέω γιατί ότι απλούστατα η βοήθεια, η ενίσχυση που δίνουμε δεν έχει λόγο αυθύπαρκτο. Δεν είναι αυτός ο σκοπός. Στόχο έχει να βοηθήσουν ανθρώπους αυτούς να σταθούν στα πόδια τους, να αναπτυχθούν οι οικονομίες τους και να μπορέσουν να λειτουργήσουν αυτόνομα. Όλα αυτά λοιπόν, αυτό το στόχο έχουν. Άρα λοιπόν, αν μπορούμε τέσσερα κράτη της Αφρικής, όπως είχαν αναλάβει και τα καθήκοντα ως Επίτροπος Αρμόδια για το Εμπόριο, να αναπτύξουμε τι δυνατότητε του για αμοιβέ μεταξύ του σχέσει, τότε ναι, γιατί τότε κράτη, Φερρυπίν, κεντρικά τη κεντρική Αφρική που ε, ε, είναι υπηρετικά, δεν έχουν πρόσβαση στη θάλασσα, μπορούν να οργανωθούν, να στείλουν τα προϊόντα του μέχρι τα λιμάνια και να τα διακινήσουν ανά τον κόσμο και να αναπτυχθούν έτσι. Δεν ε, μα προσελκύουν εμά μόνο εμπορικέ συμφωνίε. Είναι σημαντικέ οι εμπορικέ συμφωνίε, ωστόσο. Γιατί έχουμε και εμεί στι χώρε μα κάποια ζητήματα οικονομικά που πρέπει να αντιμετωπίσουμε και ω εκ τούτου το ελεύθερο εμπόριο έχει μεγάλη σημασία για μα, αλλά για τι χώρε αυτέ επίση είναι πολύ σημαντικό, γιατί προσπαθούν να χτίσουν, να οικοδομήσουν τι οικονομίε του. Και αυτό βεβαίω έχει να κάνει και με τη βοήθεια που θα προσφέρουμε, που θα είναι είτε στι υποδομέ που ανέφερα νωρίτερα, είτε στην πρόσβαση για τι αγορέ ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα δεν είναι ότι δεν είναι ανοιχτέ οι αγορέ μα, αλλά ότι αυτέ οι χώρε δεν ικανοποιούν τι προδιαγραφέ που έχουμε ορίσει. Οι δε προδιαγραφέ στόχο έχουν την προστασία του καταναλωτή, δημόσια υγεία και το καθεξή, υγιεινή και για πολλού άλλου αντίστοιχου λόγου. Άρα ναι, πολύ σωστό είναι αυτό που λέτε για την οικονομική αλλαγή μπορεί να επιφέρει πρόσβαση στις αγορές για τις λιγότερο επιτυχμένες χώρες και λιγότερα τις οικονομίες τους. Και πρόσφατα είχα συνάντηση με τις χώρες Καραϊβικής ομαδών ώστε να συζητήσουμε το πιο αποτελεσματικό τρόπο για αναζωγόνηση των των οικονομιών του και του εμπορίου τους. Ε, έμεναν πολλέ δυσκολίε για τι χώρε αυτέ όταν έγινε συζήτηση. Αυτό ακριβώ είναι και ο λόγος των οποίων από αυτέ τι πολιτικέ. Και σχετικό με αυτό είναι ότι δεν υπάρχει αμφιβολία πω όταν περνάει μέσα από μια περίοδο αστάθεια μια χώρα δεν είναι πολλές, δεν είναι λίγα τα όρο μέσα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και πάνω από όλα. Βέβαια το μέσο σταθεροποίηση που μα επιτρέπει σε σχέση με κάποια χώρα που το έχει ανάγκη να αναπτύξουμε ε, δράσεις και για την ανάπτυξη, λαμβάνοντας υπόψη βέβαια και τις πτυχές μιας ενδεχομένης περιβαλλοντικής καταστροφής. Φερρυπίν, η Ιαπωνία. Όταν πήγα τον Νοέμβριο, πήγα στη Φουκουσίμα να δω τις συνέπειες αυτού του καταστροφικού τσουσάμι. Ήταν μια από τις τσουνάμι, ήταν μια από τις πιο καταστροφικές εμπειρίες, πιο δραματικές εμπειρίες που έχω ζήσει. Έχουμε ανθρώπους που ζουν ακόμη σε πρόσκαιρα καταλήματα και βεβαίως και πρέπει να ε, γνωρίζουν και γνωρίζουν όντω ότι του έχει σταθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι ήταν στο πλευρό τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εδώ μιλάμε για μια πλούσια χώρα, για μια χώρα η οποία έχει τεράστιο δυναμικό να επιλύσει αυτόνομα τα προβλήματά τη. Αλλά πάνω στην ακτογραμμή τη έκανε μια τεράστια καταστροφή αυτό το τσουμανάμι. Και ήταν πολύ σημαντικό ότι μπορέσαμε να είμαστε παρόντε και να στηρίξουμε και τι μη κυβερνητικέ οργανώσει του. Γι' αυτό λοιπόν, οτιδήποτε έχουμε να προσφέρουμε άνω τον κόσμο πρέπει να είμαστε θέσει να είμαστε παρόντε και να το προσφέρουμε σε μια περίοδο κρίσεω. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Πέντε έχουν ζητήσει το λόγο. Συν έναν έκτο θα δεχτώ αν έχουμε χρόνο. Αμάντε Κάιζερ. Και μετά δεν θα δεχτώ άλλα αιτήματα υποβολής ερωτήματος. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Σας ευχαριστούμε κυρία Άστον που ήρθατε να μας δείτε. Σας ευχαριστούμε και για τις επεξηγήσεις σας. Πρώτο ερώτημα. Ε, πολιτική ανάπτυξης και πολιτισμός. Στην ε, Σύνοδο ΑΚΕ τον Μάιο μάθαμε και εξεπλάγημεν από ε, αυτό που μάθαμε ότι ο πολιτισμός δεν είναι πλέον επιλέξιμος. Κάτι το οποίο είναι αρκετά αρνητικό κατά την άποψή μου. Ο κύριος Πίλπαλς προσπάθησε να απαντήσει ότι επικρίνεται ε, η προσπάθεια συμπερίληψης της διάστασης του πολιτισμού στην αναπτυξιακή βοήθεια από τη στιγμή που μιλούμε για χώρες εξαιρετικά φτωχέ κτλ. Δική μου άποψη είναι ότι αυτό είναι απαράδεκτο και θέλω ε, διευκρινήσεις. Ε, το ταμείο δηλαδή αυτό, ε, το χρηματοδοτικό εργαλείο δεν θα συμπεριλάβει τα θέματα του πολιτισμού. Θέλω απάντηση από αυτού παρακαλώ. Σίγουρα ε, θα υπάρξουν αντιδράσεις από πλευράς Επιτροπής μας μπορούμε να αποφασίσουμε να συμπεριλάβουμε ξανά αυτό το θέμα στην ημερήσια διάταξη. Θέλω όμως να το διαψεύσετε ή να το επιβεβαιώσετε. Ότι δηλαδή έχει κλείσει το θέμα για σας και ότι η πολιτισμική διάσταση δεν θα λαμβάνεται πλέον υπόψη στην πολιτική ε, και σε θέματα ε, αναπτυξιακής βοήθειας. Παρόλο που κατά την άποψή μας ο πολιτισμός, η κουλτούρα είναι ένα μέσο για την ανάπτυξη. Από εκεί και πέρα, ως προς το Σουδάν παρά τις προσπάθειές μας και παρά όλα όσα έχουμε κάνει για αυτή τη χώρα, η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά δύσκολη. Είναι φρικτή και στο βορρά και στο νότο και ε, υπάρχουν θέματα ανθρωπιστικά, ε, βομβαρδισμοί, όπως γνωρίζετε, αδυναμία πρόσβαση σε συγκεκριμένα σημεία, σε συγκεκριμένες ε, τοποθεσίες, περιοχές που έχουν βομβαρδιστεί. Η κατάσταση είναι επίσης εξαιρετικά δύσκολη λόγω των πολιτικών προβλημάτων που δημιουργούνται με τα θέματα του πετρελαίου και είναι και εξαιρετικά δύσκολη σε επίπεδο αναπτυξιακής βοήθειας. Μιλούσαμε λοιπόν για την συνέχιση που θα δοθεί την παρακολούθηση μετά τις εκλογές, το follow-up. Πολλά έχουν γίνει, αυτό είναι σίγουρο, αλλά δεν έχουμε μια συνολική θεώρηση. Ε, τι ακριβώς γίνεται. Με, ξέρουμε ότι χρηματοδούμε το πάνελ υψηλού επίπεδου, αλλά ποια θα είναι τα αποτελέσματα με ποιο τρόπο. Δηλαδή είναι κάπως νεφελώδης η κατάσταση. Ε, ενώ ήταν μία από τις χώρες που αποτελούσε και αποτελεί προτεραιότητά μας. Θα ήθελα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάποια στιγμή να εμβαθύνει στο θέμα αυτό Δεν είναι δυνατόν, ενώ η κατάσταση είναι τόσο δραματική εκεί, να γίνεται τόσο λίγος λόγος, αν θέλετε, για αυτό το θέμα. Ή, εμπασίπτωση εμάς να μας ενημερώνετε τόσο λίγο για το θέμα αυτό. Ευχαριστώ, κύριος Δίαθ Ντεμέρα. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω ε, την ύπατη εκπρόσωπο για την ε, παρουσία της εδώ στην Επιτροπή μας. Έχω να της απευθύνω τρεις ερωτήσεις που αποτελούν και τρία σήματα συναγερμού ταυτοχρόνως. 13 εκατομμύρια φτωχούς έχουμε στην Ευρώπη και 75 εκατομμύρια ανθρώπους στην Ευρώπη οι οποίοι υποσυτίζονται. Από ό,τι όμως φαίνεται η πλειονότητα των φτωχών εδώ στην Ευρώπη είναι οι φτωχοί που έρχονται από εκείνες τις τρίτες χώρες. Και τι κάνει το Συμβούλιο. Θέλει να τελειώσει με τις τράπεζες τροφίμων και ε, να πάρει 500 ε, εκατομμύρια ευρώ τα οποία είναι απαραίτητα για να ε, προστατευτούν και να βοηθηθούν αυτά τα θύματα της φτώχειας και θέλει ε, να αφήσει το θέμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε επίπεδο έκφρασης αλληλεγγύης τρόπος του λέγει. Από εκεί και πέρα, έχουμε ελεύθερη κυκλοφορία ατόμων, ελεύθερη διακίνηση κεφαλαίων, προσφορά υπηρεσιών και το καθεξής, υποτίθεται. Και έρχεται η Αραβική Άνοιξη και αλλάζουμε το σημείο εστίασης, αν θέλετε, την οπτική μας γωνία και αναστέλλεται το Σέγγεν, αναστέλλεται μία από τις θεμελιώδεις ελευθερίες μας, η ελευθερία της ε, διέλευσης, ε, ε, με τα γνωστά επιχειρήματα. Εδώ όμως μόνο 13.000 έφτασαν τελικά. Πολύ μικρός αριθμός για να τεκμηριωθεί ανάγκη αναστολής μιας τόσο θεμελιώδους ελευθερίας μας. Και από εκεί και πέρα, ε, σε σχέση με αυτό που είπε και η κυρία Κέλλερ, η αναπτυξιακή, η αναπτυξιακή βοήθεια και ο έλεγχος της μετανάστευσης, δηλαδή ο έλεγχος των συνόρων. Σε ορισμένες χώρες ε, ε, χρησιμοποιείται η αναπτυξιακή βοήθεια ως μέσο ελέγχου των σύνορων για να αποφευθεί να φύγουν αυτοί οι άνθρωποι από τα ε, σύνορα. Αυτό το οποίο, για το οποίο μιλάω μεταφράζεται σε πλοία, σε αεροσκάφη, σε οχήματα 4x4 στη Σενεγάλη, στο Μάλι, στη Μαυριτανία. Είναι γνωστό αυτό και θα ήθελα την αντίδρασή σας και την απάντησή σας σε αυτές τις τρεις ερωτήσεις. Ευχαριστώ κύριε Θεοχάρους. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, ένα ερώτημα που έχω να υποβάλω ο Βαρόνι Άστον είναι ανάλογο με το ερώτημα που έχει θέσει προηγουμένως ο συνάδελφος. Χαίρομαι βεβαίως πάρα πολύ που έχει γίνει αντιληπτό, έχει γίνει πολιτική ότι η αναπτυξιακή βοήθεια είναι πιο αποτελεσματική όταν χορηγείται στο επίπεδο της κοινότητας και όχι στο επίπεδο των ε, κυβερνήσεων και πιστεύω ακόμη ότι είμαστε όλοι αφοσιωμένοι στο ζήτημα τη ε, καταπολέμησης της Ωστόσο, θα ήθελα να σα ρωτήσω τι απάντηση δίνουμε, Βαρόνι Άστον, στα εκατομμύρια, δεν είναι 13 μόνο, είναι πολύ περισσότερα, τα εκατομμύρια των Ευρωπαίων που ζουν κοντά στο όριο της φτώχειας ή κάτω από το όριο της φτώχειας, την ίδια στιγμή που βλέπουμε ότι δισεκατομμύρια, αυτά το ρωτάω με την αρμοδιότητα σας ως, ας μου επιτραπεί, έχοντας περισσότερες αρμοδιότητες σε ζητήματα και εξωτερικής πολιτικής και ασφάλειας από ό,τι αφορούσε το στενό όριο της Επιτροπής ΔΕΒΕ. Τι απάντηση δίνουμε σε αυτούς τους ανθρώπους τη στιγμή που βλέπουμε δισεκατομμύρια να ξοδεύονται είτε για να κάνουν κάποιοι ηγεμονική πολιτική στη γειτονιά τους, είτε για εξοπλισμούς, δεν θέλω να πάρω το παράδειγμα της Αργεντίνας που είπε ο, ο συνάδελφος Σοντέβα, αλλά θα μπορούσε να το σκεφτεί κάποιος και αυτό, είτε να βλέπουν να είναι τόσο αναποτελεσματική η βοήθεια και να δίνεται τόσο πολύ χωρίς έλεγχο. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Γκερέρο Ισάλομ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Να καθησυχάσω την κυρία Στρίφλερ, να σας πω ότι δεν πρόκειται να ε, χρησιμοποιήσω τα δύο λεπτά που μου έχετε δώσει, πολύ λιγότερο. Και να καθησυχάσω τον κύριο Ντέβα και την κυρία Άστον, γιατί δεν πρόκειται να παρεύω σε αυτή την αγγλοβρετανική συζήτηση για τις νήσους Φόκλαντς, οι οποίες ως γνωστόν είναι οι Μαλβίνες νήσοι. Θέλω να θέσω ένα ερώτημα για το κέρας της Αφρικής. Ε, το έχουμε δει και σε άλλες περιοχές του κόσμου. Σε περιόδους μεγάλης ξηρασίας, έχουμε δει σε περίοδο μεγάλης ξηριασίας τεράστια προβλήματα για τον τοπικό πληθυσμό. Ε, με την αλλαγή του κλίματος θα οξύνεται ακόμα περισσότερο αυτό το ε, πρόβλημα. Άρα χρειάζεται πρόληψη να μπορέσουμε εγκαίρως να ανταποκριθούμε ε, σε αυτά τα οξία προβλήματα. Θα χρειαστεί ανθρωπιστική βοήθεια μετά από αυτές τις φρικτές περιόδους ξηρασίας που έχουν παρατηρηθεί ε, στο κέρας της Αφρικής. Ε, πώς ε, θα έχουμε τα συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης για να προλάβουμε αυτά τα φαινόμενα που εμφανίζονται μετά από περιόδους έντονης εξηρασίας. Και επίσης, ε, σε σχέση με το, τις αγορές παραγόγων, έχει εγκριθεί κανονισμός ε, ούτως και πώς θα επηρεάσει αυτό την πρόληψη της κερδοσκοπίας πάνω στις τιμές των βασικών τροφίμων, βασικών πρώτων υλών. Πράγματα δηλαδή που επηρεάζουν την καθημερινότητα των πληθυσμών στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες. Πώς θα εφαρμοστεί αυτός ο κανονισμός έτσι ώστε να επηρεάσει και την αγορά των παραγωγών όπου πολλούνται τα τρόφιμα και έχουν, έχουμε τις βασικές τιμές τους που διακυμένονται. Ευχαριστώ. Ο επόμενος ομιλητής. Ευχαριστώ πολύ. Χαίρομαι που μπορώ να μιλήσω Ολλανδικά, ενώ άλλοι συνάδελφοι δυστυχώς δεν μπορούν να μιλήσουν τη γλώσσα τους. Είναι η δεύτερη φορά που έρχεστε, Βαρόνι Άστον. Είναι δυστυχές αυτό. Ε, πρέπει να είστε παρούσα, πρέπει να σας βλέπουμε πιο συχνά στη δική μας Επιτροπή. Ε, ε, επίσης ακούω ένα σωρό αρτικόλεξα και ακρονίμια τα οποία δεν πολύ καταλαβαίνω. Έχω δύο συγκεκριμένες πολιτικές ερωτήσεις να σας απευθύνω. Πρώτο για τη Λευκορωσία. Το έχετε θίξει βέβαια το θέμα. Από τη στιγμή που είναι η δεύτερη φορά που αναφέρεστε σε διπλωμάτες μιας χώρας λογικό είναι να επιμείνω. Ο Λουκασέγκο είπε και σήμερα το πρωί μάλιστα ότι η Ένωση ακολούθησε μία άγουσα, επέλεξε μία οδό κλιμάκωσης. Ποιες κυρώσεις μπορείτε να πάρετε, ε, τι μπορεί να γίνει. Φαντάζομαι ότι ενδεχομένως θα πρέπει να ληφθούν μέτρα. Όσοι στηρίζουν αυτό το καθεστώς οι υπάλληλοι ενδεχομένως μπορούν να θεωρηθούν και ένοχοι, έτσι δεν είναι. Δεύτερον, για το Ιράν. Έχει, έχετε απευθύνει έκκληση μαζί με τις Ηνωμένε Πολιτείε έτσι ώστε το Ιράν να παρετηθεί ε, της, ε, του δικαιώματος του να μην, της θανατικής ποινής, δηλαδή να, μην την εφαρμόζει πια. Ε, ποια άλλα μέτρα μπορείτε να πάρετε, όχι απλά να απευθύνετε εκκλήσεις έτσι ώστε αυτή η φρικτή κατάσταση, εν πάση περιπτώσει, να σταματήσει και να σωθούν οι ζωέ των ανθρώπων. Ευχαριστούμε. Κύριε Γκέρενς, θα είστε ο τελευταίο ερωτών. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Έχετε, έχω δύο ερωτήσει να θέσω στη Lady Διάστον. Πρώτον, σε σχέση με την απάντηση που μου δώσατε, λέει Άστον, για τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσε να συμμετάσχει περισσότερο το Συμβούλιο, με τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσαμε να εμπλέξουμε περισσότερο το Συμβούλιο και πώς ε, ε, αντιμετωπίζετε την Επιτροπή μας ε, στην υπηρεσία σας. Νομίζω ότι υπάρχει πραγματικό πρόβλημα, εκτός και αν κανείς δεν έχει σωστή αντίληψη της κατάστασης. Θέλω να υποβάλω αυτή την πρόταση. είναι βασικό μέσο. Θα πρέπει να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε πιο γρήγορα, να προχωρήσουμε πιο γρήγορα, να δεσμευτείτε για, τις, για την πρότασή μου. Αυτό καταρχάς. Κατά δεύτερο, ως προς το εμπόριο. Η προώθηση του εμπορίου παγκοσμίως ε, είναι πηγή πηγή πλούτου και μάλιστα τεράστιου πλούτου, αλλά αυτός ο πλούτος δεν κατευθύνεται εκεί που θα ήταν χρήσιμος. Στην παρουσίασή σας μιλήσατε για ένα σωρό θέματα, αλλά δεν μιλήσατε καθόλου για το εμπόριο. Είναι αδύνατο να περιλάβουμε τις οικονομικές πτυχές, τις εξωτερικές οικονομικές πτυχές, Δηλαδή στην εξωτερική πολιτική της ε- Ένωσης να περιλάβουμε τις εμπορικές πτυχές και τις οικονομικές πτυχές. Και εκεί αυτό είναι ένα μείον, ένα μειονέκτημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, στη συνθήκη προβλέπονται βεβαίως και ε, προβλέπονται ευρείες αρμοδιαιότητες. Θα πρέπει να υπάρχει περισσότερο συντονισμός και να διεξαχθεί ειλικρινής διάλογος για τα θέματα αυτά. Θα ήθελα λοιπόν να το σχολιάσετε αυτό. Όταν ήσασταν ε, επίτροπος ε, με χαρτοφυλάκια τα θέματα του εμπορίου, νομίζω ότι είχατε γνώση. Νομίζω ότι μπορείτε να τα σχολιάσετε αυτά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ να δώσω το λόγο στη Άστον, η οποία θα απαντήσει. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Ντεκάιζερ, συμφωνώ μαζί σας. Όντως το θέμα του πολιτισμού είναι πολύ σημαντικό και μάλιστα ε, για πολλούς λίγου, η κουλτούρα εκφράζει τους, τους συγκεκριμένους λαούς βεβαίως. Ε, η δυνατότητα να μπορέσουμε να υποστηρίξουμε τον πολιτισμό τους είναι κάτι που θα τους βοηθήσει εξαιρετικά να αναλάβουν δεσμεύσεις, να είναι δραστήριοι πολίτες στην κοινωνία στην οποία θα διαβιούν. Έχουμε στοιχεία εδώ και πάρα πολλά χρόνια, τα οποία αποδεικνύουν ότι κάθε φορά που κάποιος είναι περήφανος και βλέπει ότι η κουλτούρα του ε, γίνεται αντικείμενο σεβασμού, τη χάνει στήριξη, τότε ο ίδιος είναι και περισσότερο επιτυχημένος. Και όλα αυτά είναι πολύ λογικά. Ε, ε, ο Άντερς και εγώ έχουμε ε, δουλέψει πάνω σε αυτά τα θέματα. Δεν διαγράφουμε τον πολιτισμό, το βάζουμε μέσα στο μείγμα πολιτικής που προσπαθούμε να φτιάξουμε. Ε, και κάθε φορά που επισκέφτομαι ε, διάφορες περιοχές του κόσμου όπου έχουμε προγράμματα και έργα, τη βλέπω τη διάσταση του πολιτισμού. Στην Ινδία, για παράδειγμα. Δεύτερον, η βιομηχανία πολιτισμού αυτή καθεαυτή είναι ένας πολύ σημαντικός τρόπος, ένα εργαλείο για να αναπτύξει ένας λαός την ταυτότητα αλλά και την οικονομία του στη συνέχεια και μέσω της κουλτούρας και του πολιτισμού όλες οι χώρες, η κάθε χώρα του κόσμου μπορεί να αποκτήσει ιδιαίτερη σημασία. Στην Ινδία, για παράδειγμα, ε, την χάνουν στήριξη καλλιτέχνες από διαφορετικές περιοχές που ανήκουν και σε μειονοτικές εθνοτικές ομάδες. Αναγνωρίζεται, χαρτογραφείται η κουλτούρα τους, ε, ταυτοποιείται καταγράφεται και μπορούν να αναγνωριστούν με τη συγκεκριμένη πολιτιστική ταυτότητα. Και επίσης ήταν ευκαιρία να ανακαλύψουμε θαυμάσιους καλλιτέχνες, οι οποίοι θα λάμψουν στο μέλλον και έτσι θα δημιουργηθούν και ευκαιρίες ευημερία για τους λαούς αυτούς. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι που υποδεικνύει ότι ε, παραγνωρίζουμε την κουλτούρα ή την αφήνουμε στο περιθώριο. Τώρα για τον Νότιο Σουδάν. Είναι μια ε, χώρα πάρα πολύ ε, ευπαθή, συμφωνώ μαζί σας και μιλούσα και με τον την αρμόδια ε, εκπρόσωπο των Ηνωμένων Εθνών. Έχουμε και εμείς ειδικό απεσταλμένο και μίλησα με αυτούς ε, για το τι συνέβη στο Μπρουνάλ αλλά και στο Νταρφούρ. Νομίζω ότι ε, γίνεται προσπάθεια να γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ Βορρά και Νότου, να λυθεί το θέμα των συνόρων, το θέμα των αγωγών και να μειωθούν τα προβλήματα στις αμφιλεγόμενες περιοχές είναι σημαντικό να γίνει μεγάλη προσπάθεια και μάλιστα διεθνής προσπάθεια και θα συνεχίσουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Και μάλιστα και πολλά χρήματα αφιερώνουμε σε αυτό. Ε, ε προσπαθώ να βρω τα στοιχεία. Αν δεν απατώμε, μιλούμε για 700 εκατομμύρια ε, ευρώ για τα επόμενα χρόνια συνολικά. Και γι' αυτό προσπαθούμε να φτιάξουμε υποδομέ. Μίλησα, ε, ανέφερα προηγουμένω και το αεροδρόμιο, κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό γιατί γενικά το ταξίδι, η μετακίνηση, οι μεταφορές στη χώρα αυτή είναι πολύ προβληματικέ. Και η εξέβρεση λύση ε, για το θέμα του αγωγού και των αγών θα είναι πραγματικά πολύ σημαντική. Ελπίζω ότι οι συσκέψεις που βρίσκονται εν εξελίξη θα οδηγήσουν στην επίλυση αυτού του προβλήματος. Έτσι ώστε τελικά η οικονομία στο Νότο να ε, μπορέσει να επωφεληθεί ε, από ε, το, τις πετρελαϊκές πηγές και αυτή του Βορρά να επωφεληθεί από την ε, μεταφορά του πετρελαίου. Βεβαίως, εμείς λέμε συνεχώς ότι δεν μπορούμε να καλύψουμε το κενό που θα δημιουργηθεί από την απώλεια αυτού της, της τεράστιας πηγής εισοδήματος. Θα πρέπει να βρεθεί μια συνολική ουσιαστική λύση. Ε, τώρα, κύριε Δίας Δεμέρα, μιλήσατε για μια, αναφέρατε μια σειρά προβλημάτων ε, εσωτερικών. Ένα από τα πράγματα που έχουν μεγάλη σημασία στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι το εξής. Είμαστε σε θέση να αναγνωρίσουμε πόσο σημαντικά είναι τα δικά μας κεκτημένα και θέλουμε να δείξουμε στις άλλες χώρες τα ωφέλη που έχουμε να τους προσφέρουμε. Για παράδειγμα, η ελεύθερη κυκλοφορία των ατόμων. Ε, να σας δώσω ένα παράδειγμα. Πιστεύω δύο πράγματα. Οι φοιτητέ, οι επιχειρηματίε, όλοι οι άνθρωποι, όσο περισσότερη στήριξη έχουν, όσο περισσότερε δυνατότητε του δίνονται να σπουδάζουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή να έρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση για επιχειρηματικού λόγου, για δουλειέ, τόσο ε, ε, ε, πιο ωφελημένη θα βγει η σχέση μας, η αμοιβαία σχέση μας με τις χώρες προέλευσής τους, γιατί έτσι επιστρέφοντας στη χώρα τους θα ε, θα αναζωπυρώσουν την οικονομία και θα την ε, κάνουν τη χώρα πολύ πιο σύγχρονη, με την οποία ε, θα συνεργαστούμε και καλύτερα στο μέλλον. Αυτό καταρχάς. Ε, κατά δεύτερο λόγο, συνήθως όντως οι, οι άνθρωποι προτιμούν να μένουν στην πατρίδα τους και να συμμετάσχουν στην αναπτυξιακή προσπάθεια της πατρίδας τους. Σε όλα τα μέρη που έχω πάει, βλέπω ότι γενικά η πλειοψηφία θέλει να μείνει στη χώρα αυτή και αναγκάζεται να φύγει και να έρθει ενδεχομένως προς τα εδώ δεν έχει προοπτικές εκεί. Όσο περισσότερο τους στηρίζουμε επί τόπου να παραμείνουν με τους φίλους τους, με τις οικογένειές τους, τόσο το καλύτερο για όλους. Και οι πολι... όλες αυτές οι πολιτικές πρέπει να ενταχθούν σε αυτό το ευρωπαϊκό καλάθι αξιών και ε, ε, ιδεών ε, τις οποίες εμείς ενστερνιζόμαστε και οι οποίες είναι τόσο σημαντικές για εμάς. Τώρα, κυρία Θεοχάρους, για το... ως προς το θέμα της αναπτυξιακής βοήθειας και της αξίας αυτής, Πώς έχουμε δηλαδή πραγματική αξία από την αναπτυξιακή βοήθεια. Ναι, αυτό είναι μία από τις ε, πιο ε, μεγάλες προκλήσεις για μας. Πρέπει να βρούμε πιο έξυπνους τρόπους αντίληψης του ε, αντικτύπου που έχει η αναπτυξιακή μας βοήθεια. Αν εξετάζουμε τα αναπτυξιακά θέματα ξεχωριστά, τότε χάνουμε τη δυναμική ε, την, ε, που μας προσφέρει το σύνολο των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το εμπόριο, η εφόρος ανάπτυξη, η δουλειά που κάνουμε για τις κλιματολογικές αλλαγές, ο τρόπος με τον οποίο στηρίζουμε τους πληθυσμούς σε περιπτώσεις κρίσεων, ε, τι κάνουμε για να ενισχύσουμε τη σταθερότητα του, πολιτικού καθεστώτος σε κάθε χώρα, τα, η δράση μας για το περιβάλλον. Όλα αυτά πρέπει να ε, ταιριάζουν μεταξύ τους. Όλες οι ευρωπαϊκές πολιτικές θα πρέπει να κατευθύνονται προς την ίδια κατεύθυνση, να κατευθύνονται προς τον ίδιο δρόμο, ούτως ώστε να είμαστε αποτελεσματικοί, να έχουμε ε, σωστή σχέση αξίας προς τιμή, να μπορέσουμε πραγματικά να αλλάξουμε τις ζωές των ανθρώπων. και πρέπει βεβαίως να δούμε πώς η πολιτική μας επηρεάζει τις πιο ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, πώς βοηθούμε τους ανθρώπους τελικά να αξιοποιήσουν όλες τις δυνατότητές τους και πώς μπορούμε να τους βοηθήσουμε να αποκτήσουν τον έλεγχο της ζωής τους, της κοινωνίας τους, να αναλάβουν δηλαδή ευθύνες περισσότερες όσο περισσότερη συνοχή έχουμε στη δράση μας, τόσο περισσότερο μπορούμε να μετρήσουμε, να αξιολογήσουμε τη δράση μας, να δούμε κατά πόσο πιάνουν τόπο, δηλαδή, αν θέλετε, τα χρήματά μας. Και πάντοτε στο επίκεντρο των δράσεών μας πρέπει να είναι οι ευρωπαϊκές αξίες. Κύριε Κερερό, αναφερθήκατε στο συγκεκριμένο πρόβλημα της ξηρασίας και των συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης έναντι των λιμών μετά την ξηρασία. Βεβαίως, ε, ε, από τη μία έχουμε έναν τεράστιο όγκο πληροφοριών που περιγράφει τι αντίκτυπο θα έχει η αλλαγή του κλίματος σε πάρα πολλές χώρες. Τουλάχιστον 100, αν όχι και παραπάνω χώρες, θα πληγούν ιδιαιτέρως ε, και θα είναι εξαιρετικά ευπαθείς λόγω των αλλαγών του κλίματος. Σε κάποιες, κάποιες θα υποστούν εξαιρετικά μεγάλες πλημμύρες και κάποιες εξαιρετικά μεγάλες περιόδους ξηρασίας. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε γενικότερα είναι το εξής. Ε, όλες οι υπηρεσίες ε, συνεργάζονται για να έχουμε στήριξη εγκαίρως, να προσφέρουμε στήριξη εγκαίρως, να ενημερώσουμε εγκαίρως τις χώρες, να δούμε τι μπορούμε να τους προσφέρουμε στο επίπεδο της, της βοήθειας, ελπίζοντας ότι ο πληθυσμός θα παραμείνει επιτόπου. Έχουμε δει όλες τις τηλεοράσεις μας και γνωρίζουμε ότι τι ακριβώς γίνεται και κάνουμε και συζητήσεις στις χώρες μας και ξέρουμε ότι όλα αυτά είναι φιλοδοξία, δεν υλοποιούνται πάντοτε. Πολλές περιοχές που πλήττονται από ξηρασία είναι και περιοχές όπου έχουν ξεσπάσει συγκρούσεις και χρειάζεται πολύ μεγαλύτερη προσπάθεια και χρειάζεται πολύ μεγαλύτερη στήριξη. Νομίζω ότι ε, έχουμε λοιμούς αυτή τη στιγμή, τους οποίους πρέπει να αντιμετωπίσουμε και θα πρέπει να προσφέρουμε περαιτέρω στήριξη. Χρειάζεται να έχουμε πιο μακροπρόθεσμες προβλέψεις, έτσι ώστε να εξετάσουμε πώς η αλλαγή του κλίματος θα επηρεάσει ε, και την ε, επισητιστική αν θέλετε επάρκεια, την επάρκεια των τροφίμων, την ασφάλεια στην προμήθεια των τροφίμων, την ασφάλεια στους υδάτινους πόρους, την αποθήκευση αυτών, στη χρήση όλων αυτών. Ε, τι επιπτώσεις δηλαδή θα έχει ε, στον γενικότερο τομέα των τροφίμων η αλλαγή του κλίματος. Να δούμε ε, ποιες αλλαγές δηλαδή θα υποστεί το, το μοντέλο αυτό, ούτως ώστε να μπορέσουμε να προβλέψουμε. Θα έλεγα ότι το νερό, η υδάτινη πορή είναι ένα αγαθό τόσο σημαντικό που πραγματικά θα δώσει λαβή και ήδη δίνει λαβή για πολύ έντονες συγκρούσεις και αυτό θα γίνει πολύ πιο έντονο στο μέλλον. Τώρα, ε, πώς θα επηρεάσει η δράση μας ευνοϊκά ε, την αγορά των παραγόγων δεν το γνωρίζω ακόμα, αλλά θα, θα το διερευνήσω και θα επανέλθω να σας απαντήσω πιο συγκεκριμένα. Τώρα, ε, να απαντήσω στον ομιλητή που μου, μου έθεσε ερωτήσεις για την Λευκορωσία και το Ιράν. Έχουμε προβλέψει κυρώσεις για την Λευκορωσία, πρέπει να επανεξετάσουμε το καθεστώς των κυρώσεών μας, έτσι ώστε να είμαστε σίγουροι ότι είναι αποτελεσματικές οι κυρώσεις, ότι ασκούν πίεση και να δούμε και με ποιο τρόπο μπορούμε άλλωστε να τα αποφύγουμε όλα αυτά για να πετύχουμε αυτό που πραγματικά θέλουμε. Έχετε δίκιο στην παρατήρησή σας ε, είναι καλό να, είμαστε, να έχουμε στοχευμένη προσέγγιση, να έχουμε μια ε, στοχοπροσύλωση και αυτό προσπαθούμε να το κάνουμε και στην περίπτωση της Λευκορωσίας, μεταξύ άλλων. Πάντοτε στόχος μας είναι να ε, επικεντρωθούμε σε συγκεκριμένα άτομα, σε συγκεκριμένες οργανώσεις, άτομα ή οργανώσεις που μπορούν πραγματικά να επηρεάσουν το καθεστώς. Το προσπαθούμε πολύ και στο Ιράν κυρίως, αλλά και αλλού προσπαθούμε να, η δράση μας να μην ε, έχει ως στόχο τον ε, γενικότερο πληθυσμό. Είναι δύσκολο αυτό, αλλά είναι εξίσου σημαντικό. Έχετε δίκιο, η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, εργάζεται όλοι, όλα τα μέλη συνεργάζονται και προσπαθούν να ασκήσουν πίεση όλοι οι πρέσβεις στη Λευκορωσία και επομένως είναι, παράδειγμα, είναι ένα παράδειγμα καλής συνεργασίας. Τώρα, ως προς το εμπόριο, νομίζω ότι, ε, κύριε Γκέρενς, ότι πραγματικά σχολίασα τα θέματα του εμπορίου αρκετά. Το εμπόριο πρέπει να ενσωματωθεί με ξεκάθαρο τρόπο στην ε, πολιτική μας. Ε, Πρέπει να έχουμε μια στρατηγική προσέγγιση του πώς γίνεται αντιληπτή η Ευρώπη στον υπόλοιπο κόσμο. Νομίζω ότι η μέρος της εξωτερικής μας πολιτικής έχει στόχο την στήριξη των ευρωπαϊκών λαών. Ε, θέλουμε οι, ευρωπαϊκοί λαοί που πραγματικά έχουν εμπιστοσύνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση να συνεχίσουν να το κάνουν, αλλά και οι λαοί από τρίτε χώρε. Αν καταστήσουμε έναν κόσμο πιο ασφαλή, ε, για όλους, αυτό θα είναι καλό για όλους μας. Αν, μπορούμε να έχουμε καλές εμπορικές σχέσεις, ελεύθερο εμπόριο, αυτό θα ε, ωφελήσει τους πάντες. Και αυτό πρέπει να εξεταστεί ε, συνολικά. Ποια αντίληψη έχουμε για τον υπόλοιπο κόσμο, ποια είναι η προσφορά, τι μπορούμε να προσφέρουμε στον υπόλοιπο κόσμο για μένα το εμπόριο έχει καθοριστική σημασία. Εξού και ε, είχαμε την πρόσφατη ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το εμπόριο και την ανάπτυξη. Ευχαριστώ. Θα τελειώσουμε τη συνάντησή μας με τη Λέδη Άστον. Σας ευχαριστούμε για το χρόνο που μας αφιερώσατε. Ελπίζω να τα ξαναπούμε σύντομα.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 Ευχαριστώ τους συνεργάτες. Να καθίσουν παρακαλώ. Θα κάνουμε ένα ηλεκτρονικό έλεγχο για την ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίστε παρακαλώ δοκιμαστικά. Λείπουν τέσσερις, λείπουν τρεις, λείπουν δύο, ένας. Εντάξει, ψήφισα και εγώ, τελειώσαμε. Καλώς λοιπόν το σύστημα λειτουργεί. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν Λοιπόν, έκθεση Κάτσμαρεκ. Τροπολογία κοντ 1. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 2 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Λοιπόν, περνάμε τώρα στην 3. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 6 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 4 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 7 υπέρ κατά 5 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 12 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 13 υπέρ κατά αποχές, ηλεκτρονικός έλεγχος για τη 13, ξεκινάει η ψηφοφορία. Ψηφίζει ένας παραπάνω. Τώρα εντάξει. Τέλος της ψηφοφορίας δεκτή. 14. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 15. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 8 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 16 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 17 υπέρ κατά αποχές δεκτή νομίζω. Ηλεκτρονικός έλεγχος παρακαλώ. Τέλος της ψηφοφορίας. Δεκτή. 18. Καταπίπτει. 16 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 8 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 9 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 10 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 19 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 20 υπέρ κατά παρακαλώ κλείστε τα τηλέφωνα δεκτή 10 υπέρ κατά δεκτή 20 11 υπέρ κατά δεκτή 22 υπέρ κατά αποχές δεκτή η ένα φετ ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές δεκτή 3, 2 μάλλον υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 3 υπέρ κατά αποχές δεκτή 4 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 5 υπέρ. Κατά αποχές έλεγχος. Λοιπόν, ψηφίζουμε την 5. Τέλος. Απορρίπτεται η 5. 6 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 7 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 8 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 9 υπέρ. Α, για μια στιγμή, σε δύο τμήματα η 9. Το πρώτο τμήμα ποιο είναι υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος για το πρώτο τμήμα της 9 παρακαλώ, ψηφίζεται. Τέλος. Υπέρ, δεκτή. Λοιπόν, 9 δεύτερο τμήμα, υπέρ, κατά. Αποχές απορρίπτεται. 10 υπέρ, κατά αποχές δεκτή. 11 έχει καταπέσει. Τελική ψηφοφορία, ποιοι είναι υπέρ. Α, για μια στιγμή λέει η πρόεδρος. Λοιπόν, ψηφίζουμε. Δεκτή η έκθεση. Ευχαριστούμε τον κύριο Κατσμάρεκ. Περνάμε στη δεύτερη ψηφοφορία. Μια και υπάρχει συμφωνία ανάμεσα στον εισηγητή και τον Σκιώδη για, τους δύο, για τις δύο επόμενες ψήφους, μπορούμε να ψηφίσουμε ο μπλοκ ομαδών. Λοιπόν, η επόμενη ψήφος θα περιλαμβάνει τις τρεις τροπολογίες του κ. Βέρμαν. Ποιοι είναι υπέρ κατά, αποχές, δεκτή. Τελική ψήφος, ηλεκτρονικά ψηφίζεται παρακαλώ. Τέλος, ομόφωνα δεκτή η έκθεση Μπέρμαν. Περνάμε τώρα, πάλι ο μπλοκ, εφόσον ομαδών όπως ε, λέγεται, στην επόμενη ψήφο, από την τροπολογία 1 μέχρι το τέλος. Όλες οι τροπολογίες. αν η προφορική ε, γίνεται δεκτή, τότε θα καταψηφιστεί η 6. Λοιπόν, ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Τελική ψήφος, ποιοι είναι υπέρ, ψηφίζεται. Ψηφίζει ένας παραπάνω. Λοιπόν, δεν πειράζει, ε, εν πάση περιπτώσει γίνεται δεκτή. Ομόφωνα δεκτή, συγχαρητήρια. Επόμενη ψήφος αφορά πρέντα, ε, ένα, ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, ηλεκτρονικός έλεγχος για την ένα. Πάλι ένας παραπάνω ψηφίζει. Α, όχι, δεν είναι ένας παραπάνω. Λάθος απορρίπτεται έτσι κι αλλιώς η ένα. Δύο, ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Τρία, ποιοι είναι υπέρ. Κατά. αποχέ δεκτή. Τέσσερα, ποιοι είναι υπέρ. Κατά. αποχέ απορρίπτεται. Πέντε, ποιοι είναι υπέρ. Κατά. απόχέ δεκτή. Προφορική ένα Ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. 6 καταπίπτει. Συμβιβαστική α κεφαλαίο. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 7. Ποιοι είναι υπέρ. Οι 9 μάλλον. Οι 2, οι 7 και 8 καταπίπτουν. Οι 9. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Οι 10 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 11 υπέρ. Κατά. Αποχές Απορρίπτεται. Τοπολογία 12. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος για τη 12. Πέρας ψηφοφορίας. Δεκτή. 13. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Προφορική 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Η 14 καταπίπτει, η 15 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Η παφορική 3 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Η 16 καταπίπτει, η 17 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 18 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 19 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 20 σε δύο τμήματα. Το πρώτο τμήμα, ποιοι είναι υπέρ Α, για μια στιγμή έχει καταπέσει το πρώτο τμήμα της τροπολογίας 20. Τελική ψήφος, εν πάση περιπτώσει. Ηλεκτρονικά ψηφίζεται το σύνολο. Τέλος ψηφοφορίας. Δεκτή. Συγχαρητήρια. Α, κυρία Ζανίκη, είδατε τι γρήγορα που τα λέω.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 Σας θυμίζω ότι έχουμε ακόμα δύο ψηφοφορίες. Έχουμε ακόμα, θυμίζω, δύο ψηφοφορίες. Παρακαλώ μη φεύγετε. Nous avons encore deux flèches. Λοιπόν, δύο γρήγορε ψήφου. Κάθε φορά πρόκειται για την τελική ψηφοφορία. Δεν υπάρχει καμία τροπολογία. Περιμένω και τον κύριο Γκουερέρο να καθίσει. Donc, euh, Ηλεκτρονική ψήφος και στις δύο περιπτώσεις. Καταρχάς ξεκινάμε με το σχέδιο γνωμοδότησης. Ποιοι είναι υπέρ. Ηλεκτρονικός έλεγχος λοιπόν, σχέδιο γνωμοδότησης ψηφίζεται. Λοιπόν, το δεύτερο Ψηφίζετε. Le vote est clos. Adopté. Voilà. Voilà. Δεκτές και οι δύο. Υπάρχει άλλο ένα θέμα. Μη φύγετε παρακαλώ. Είναι κρίμα να φύγετε λέει πρόεδρε. Είναι το σημείο 14. Έχουμε να κάνουμε με την παρουσίαση του κυρίου Νόιζερ που απευθύνεται στην Ήτρε σχετικά με την επένδυση στη συνεργασία με εταίρους πέραν των συνόρων μας στον τομέα της ενεργειακής πολιτικής. Στρατηγική αντιμετώπιση για προμήθεια ενέργειας με ασφαλή, διαρκή και ανταγωνιστικό τρόπο. Παρακαλώ λίγη ησυχία, έτσι ώστε ο κύριος Νόιζερ να περάσει να πάρει το λόγο. Νόιζερ, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πρόκειται για μια γνωμοδότηση της Επιτροπής μας για μια βιώσιμη πολιτική για την ενέργεια. Σε μια έκθεση στις αρχές του μήνα συζητήσαμε την ενεργειακή πολιτική για, την για τα αναπτυσσόμενα κράτη για το, η χρονική περίοδο έως το 2030. Την παρουσιάσαμε στο Κοινοβούλιο και τώρα έχουμε τη γνωμοδότηση για την Επιτροπή Ήτρε στην ίδια λίγο πολύ κατεύθυνση, απλώς πιο σύντομη. Και νομίζω ότι θα πρέπει να καλωσορίσουμε το γεγονός ότι η Επιτροπή ε, αφοσιώνεται στο στόχο της οικουμενικής, της παγκόσμιας πρόσβασης στην ενέργεια, ιδιαίτερα καθώς εορτάζουμε το έτος ε, της ενέργειας για τους πάντες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν, το Συμβούλιο, το Κοινοβούλιο, προσδιορίζουμε ο καθένα τα, τους στόχους μας, τα καθήκοντα που ορίζουμε για τον εαυτό μας και έχουμε την αναφορά του στόχου της οικουμενικής πρόσβασης για την ενέργεια. Δηλαδή ανανεώσιμες ενεργειακά αποδοτικές, μικρές, ε, μικρής κλίμακας και οικονομικές ενεργειακές λύσεις με ενισχυμένη συνεργασία στον χώρο της ε, ενέργειας μεταξύ εταίρων χωρίς την οποία δεν είναι δυνατή η ανάπτυξη. Και ιδιαίτερα στην ενεργειακή πολιτική για την ανάπτυξη πρέπει οι στόχοι οι αναπτυξιακοί να λαμβάνονται υπόψη και δι στόχοι της χρηστής διακυβέρνησης, τα ανθρώπινα δικαιώματα, η ε, πρόοδος προς τη δημοκρατία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση στις διαπραγματεύσεις της με τρίτες χώρες θα πρέπει επιτακτικά να δίδει έμφαση στα δικαιώματα των πολιτών και λιγότερο στα συμφέροντα των κυβερνήσεων. Επίσης επικεντρωνόμαστε και στη διαφάνεια, το δημοκρατικό έλεγχο, την συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών. Τέλος, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να μεριμνά ιδιαίτερα ώστε στον τομέα των βιοκαυσίμων να αποφεύγονται αρνητικά οικονομικά, περιβαλλοντικά, κοινωνικά ε, αποτελέσματα της χρήσης τους. Αυτά λοιπόν, όπως είπα, πρόκειται για τη γνωμοδότηση που απευθύνουμε στην αρμόδια ε, καθήλυν επιτροπή για την ε, ενέργεια, την έρευνα, τεχνολογία. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Νάιζερ και τώρα παρακαλώ τους συναδέλφους που θέλουν το λόγο. Η κυρία Κέλλερ πρώτα. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω, να εκπροσωπήσω πάνω την κυρία Γκρέσ, την σκιώδη συγκητριά μου στο βαθμό που μπορώ. Κατά βάση συμφωνούμε με τις προτάσεις που έχει περιλάβει η γνωμοδότηση. Το ερώτημα βέβαια είναι τι καινούριο θα μπορούσαμε να προσθέσουμε. Ξέρουμε ότι είχαμε το ένα και άλλες αποφάσεις που έχουμε λάβει, επομένως πρόκειται για μια μεγάλη πρόκληση. Ίσως κάποιες τροπολογίες ή κάποια τροπολογία για την πέμπτη παράγραφο να υποβληθεί από πλευράς μας εκεί όπου γίνεται λόγος για τα βιοκάψιμα. ώστε να επισημάνουμε τον κίνδυνο της μονοκαλλιέργειας πρέπει να τη θείο στόχο των βιοκαυσίμων που θα μπορούσε να οδηγήσει σε προβλήματα στι καλλιέργειε γενικότερα στη γεωργία και σε απώλεια πολύ σημαντικών ε, φυσικών πόρων. Καταστραφή δασών και λοιπόν περιβαλλοντικών στοιχείων. Επίσης, ως προς την ε, μαζική παραγωγή, στην βιομάζα, στην εκθεσία, πάλι, ήταν μια προφορική ερώτηση. Εν πάση περιπτώσει δεν ψηφίστηκε και ως εκ τούτου είναι ένα θέμα το οποίο θέλουμε να επαναφέρουμε. Και μια και πρέπει να κάνουμε τη γνωμοδότηση για το ΦΛΕΚΤ, θα ήταν καλό πιστεύω να πούμε δύο λόγια, να ενσωματώσουμε δύο λόγια μέσα στην γνωμοδότηση αυτή και για τη βιομάζα, που πιστεύω θα έπρεπε να προβλέπετε. Συμπλήρωση λοιπόν μόνο. Κατά τα άλλα μας ικανοποιεί η γνωμοδότηση. Και ελπίζουμε ότι θα εγκριθεί όπως έχει με τις μικρές αυτές εκκληρώσεις. Ευχαριστώ κυρία Σνίμπερ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Και ευχαριστώ τον κύριο Νόιζερ για την έκθεση, ιδιαίτερος δε για την επισήμανση του, προ... του ζητήματος της πολιτικής συνοχής συνέπειας. Γιατί πολλές φορές έχουμε την εντύπωση ότι αντίστροφα προσεγγίζουμε το πρόβλημα, ότι δηλαδή λέμε ε, περισσότερο τι μπορεί περισσότερο να προσφέρει η αναπτυξιακή πολιτική σε μια ενεργειακή πολιτική και όχι το ανάποδο. Νομίζω ότι τα ζητήματα αυτά θα πρέπει να τα συζητήσουμε περισσότερο, αλλά πάντως είμαστε πολύ ικανοποιημένοι. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα παρακαλώ την Επιτροπή, εάν έχει τον εκπρόσωπό της εδώ, να λάβει το λόγο. Οι συνάδελφοί μου είναι καθοδόν πρόεδρε, τους ειδοποίησαν να φτάσουν για τις παρατέταρτο. Η πρόεδρος. Ναι, ναι, πάντα το ίδιο πρόβλημα έχουμε όμως. Ας έχει την καλοσύνη η Επιτροπή να έρθει στην ώρα της τουλάχιστον. Μπορεί να είμαστε λίγο νωρίτερα στο πρόγραμμά μας, αλλά θα μπορούσαν να έρχονται και πέντε λεπτά. Δεν είναι παράλογο να στούμε να έρθουν πέντε λεπτά νωρίτερα. Δεν μπορούμε να καθόμαστε ένα τέταρτο να σας περιμένουμε. Δεν είναι φυσιολογικό αυτό τώρα. Θα πρέπει να προβλέπετε ότι μπορεί κανεί να προχωρήσει πιο γρήγορα στο πρόγραμμα ή να καθυστερήσει. Το ελάχιστο που έχει να κάνει η Επιτροπή είναι να έρχεται τουλάχιστον ένα τέταρτο νωρίτερα. Δεν έχουμε τελειώσει και μια ώρα πιο νωρί. Α, κάθομαι να περιμένω εγώ τώρα τρία τέταρτα τη ώρα μέχρι να φτάσει η Επιτροπή. Ο κύριο Νόιζερ. Και σα παρακαλώ να διαβιβάσετε το μήνυμα. Δεν είναι η πρώτη φορά που σημαίνει αυτό και το θεωρώ απαράδεκτο. Äh, Κύριος Νόιζερ, ευχαριστώ πολύ τις δύο συναδέλφους για τις παρατηρήσεις και τις συμπληρώσεις. Η πολιτική συνοχή δεν είναι ένα θέμα δικό σας μόνο, ένα θέμα που πρέπει να είναι πάντοτε δικό μας θέμα. Να το ενστερνιζόμαστε όλοι. Για την κυρία Κέλλερ βεβαίως ε, συμφωνώ. Θα συζητήσουμε τα θέματα που θα πρέπει εμείς ως Επιτροπή Ανάπτυξης να ενσωματώσουμε μέσα. Ευχαριστώ πολύ και πάλι. Πολύ καλά, κύριε Νόισερ, λυπούμε που δεν είναι εδώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όχι μόνο για σας, αλλά και για του συναδέλφου, για όλους τους εδώ παρόντε. Πέρα τη σα, αύριο το πρωί ξαναρχίσουμε στις 9. Και καλό σας βράδυ.